αλλά και σε κάθε άλλον τομέα. Κλείνω με αυτά, σημειώνοντας ότι χαίρομαι ιδιαίτερως για τη σημερινή ευκαιρία που μας δίνεται. Ευχαριστώ, Συντόνια. Λοιπόν, ε, ακούσαμε κάποιες ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις και είχαμε ε, τις ομιλίες αυτές για το αντικείμενο της ανταλλαγής απόψεων και είχαμε και μια παρουσίαση κατάσταση των πραγμάτων από τη μια όσον αφορά την κατάσταση ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού και τους περιορισμούς δημοσιονομικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, τις παρουσίες η Συντόνια και από την άλλη την έκθεση και την παρουσίαση ε, του οίκου Deloitte, ε, όσον, Deloitte όσον αφορά ε, την σχέση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με, τα, με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και πραγματικά αυτό έδειξε ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστούς κόσμους. Και μέχρι στιγμής όταν έπρεπε να ε, υλοποιήσουμε κοινού ευρωπαϊκού στόχου, ιδιαίτερα του στόχου που περιέχονται σε αυτό που ονομάζουμε στρατηγική τη Λισαβόνα, Υπήρξε πολύ ε, λίγο συντονισμός ε, των τεκτενομένων σε εθνικό επίπεδο και των τεκτενομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2000 στη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχικοί Κρατών Κυβερνήσεων αποφάσισαν ε, ε, να θέσουν μέχρι το 2010 το φιλόδοξο στόχο η ε, ε, ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, θέτοντα ορισμένε προτεραιότητε στον τομέα τη έρευνα, τη καινοτομία, ε, των νέων τεχνολογιών, της οικονομία, τη γνώση, μέσω της ανάπτυξης της επαγγελματική κατάρτιση, της εκπαίδευση κτλ. Η υλοποίηση αυτών των στόχων κατά 80% ε, αφορούσε εθνικέ αρμοδιότητε και όχι ευρωπαϊκή κοινωνική αρμοδιότητα. Άρα χρηματοδότησε από του εθνικού υπερπολογισμού. Στην πράξη, όπω έδειξε και η μελέτη ε, ε, που ανέλησε τέσσερι τουλάχιστον χώρε από τον Νίκο Ντελόιτ, η εθνική λοιπόν δημοσιονομική πολιτική δεν έλαβε πραγματικά υπόψη ε, τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Και να λοιπόν φτάσαμε ε, στο 2010 και φιλο... ο φιλόδοξο στόχο ε, τη Λισαβόνα δεν εκπληρώθηκε και η στρατηγική απέτυχε. Σε 15 ημέρε, ε, περίπου ε, θα επαναληφθεί αυτή η άσκηση πλέον με, με, με ε, ορίζοντα ε, την Ευρώπη το 2020 με στόχο εξυγίανση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών, έξοδος από την κρίση και μεσοπρόθεσμα ε, κινητοποίηση των δυνάμεων έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας το 2020. Αν θέλουμε λοιπόν αυτή τη φορά το εγχείρημα να στεφτεί από επιτυχία, σίγουρα πρέπει να εργαστούμε με διαφορετικό τρόπο. Και η πεποίθηση δική μου είναι ότι θα πρέπει Μεταξύ των άλλων, τα κοινοβούλια, τα εθνικά κοινοβούλια συνεργαστούν πολύ περισσότερο και μεταξύ του και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, με βάση αυτά, δίνουμε ε, το λόγο σε εσά. Ανάμεσα στις ε, χώρες που εκπροσωπούνται, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω ιδιαίτερα την αντιπροσωπεία του Bundestag, που ε, ήρθε ασυνήθιστα πολύ άριθμη θα λέγαμε. Γιατί είπαμε όχι πάνω από τέσσερα άτομα ανά αντιπροσωπεία, ανά κοινοβούλιο, αλλά με ε, κατά ευτυχή συγκυρία το Bundestag ε, εκπροσωπείται σήμερα στις Βρυξέλλες από πολλά μέλη ε, του κοινοβουλίου αυτού που συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές. Έξι λοιπόν είναι οι εκπρόσωποι του Bundestag και ε, κυρίως ε, χαιρετίζω τον, κύριο, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού, Επιτροπή που ασχολείται με ευρωπαϊκά θέματα. Θα αναγκαστεί να φύγει στις 4.30 για να πάει σε μια άλλη συνεδρίαση. Αν ο κύριος Χάκμαν ή κάποιο άλλο μέλος του Bundestag θέλει να πάρει το λόγο, σας παρακαλώ, μιλήστε τώρα για να μπορέσουμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε την παρουσία τους. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για, την, ε, για το χαιρετισμό σας και ε, ε, τα καλά λόγια που αναφέρατε για την αντιπροσωπεία μας και ε, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας όπως δείξατε και εσείς και τους συναδέλφους με την αντιπρόεδρο μιας άλλης ομάδας δηλαδή πώς μπορεί να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την εκτελεστική εξουσία και να εκπονούμε προτάσεις, ίσως σε ομάδες εργασίας. Είναι μία πρόταση την οποία πρέπει να ε, εμβαθύνουμε ε, για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε και ε, να την εφαρμόσουμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή, καλή επιτυχία στις εργασίες αυτής της συνεδριάσεως. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Μου κάνετε ένα ερώτημα και εφόσον θα φύγετε αρκετά γρήγορα θα απαντήσω αμέσως πράγμα το οποίο θα επιτρέψει ίσως στους άλλους ομιλητές να αντιδράσουν στην πρόταση την οποία θα διατυπώσω. Λοιπόν, το θέμα που τίθεται είναι πώς μπορούμε συγκεκριμένα να καταρτήσουμε από κοινού μία μέθοδο εργασίας που θα μας επιτρέπει να εργαζόμαστε πιο τακτικά και πιο αποτελεσματικά από μία συνεδρία στο χρόνο όπως συνηθίζεται τώρα. Εγώ θέλω να θέσω μία ιδέα προς συζήτηση. Είδατε πριν από λίγες μέρες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πρότεινε για να υπάρξει καλύτερο συντονισμός των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλει στις Βρυξέλλες το προσχέδιο του προπολογισμού ε, ώστε να εξεταστεί από τους Υπουργούς Οικονομικών και τις Ευρωπαϊκές Αρχές και αν εμφανίζεται συμβατός με τις κοινοτικές αρχές θα επιτραπεί στο Κοινοβούλιο στη συνέχεια να προβεί στην υποβολή του σχεδίου προπολογισμού στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η ιδέα μου. Νομίζω ότι ορισμένοι θα έχουν αντιρρήσεις διότι έχω ήδη, ακούσει αρνητικά σχόλια ήμουν ε, Υπουργό επί του προϋπολογισμού στη Γαλλία και δεν νομίζω ότι ο ομόλογός μου αυτή τη στιγμή πρόκειται να ε, αποδεχθεί έναν τέτοιο προκατακτικό έλεγχο αλλά προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα οι, τα κοινοβούλια να συμμετέχουν καταρχήν σε αυτό το συντονισμό. Διότι στα περισσότερα κοινοβούλια έγινε μια συζήτηση τον οποίο ονομάζουμε στη Γαλλία δημοσιονομικού προσανατολισμού σχετικά με ε, ε, την κατεύθυνση του προπολογισμού. Δεν υπάρχει παντού το ίδιο οικονομικό έτος και δημοσιονομικό έτος γιατί ε, σε άλλες χώρες είναι Ιανουάριος ως Δεκέμβριος και σε άλλες όχι. Οπότε στην αρχή της περίοδου το φθινόπωρο υποβάλλεται το σχέδιο το οποίο ε, τελικά ψηφίζεται το φθινόπερο. Τουλάχιστον έτσι κάνουμε ε, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οπότε γιατί να μην συμφωνήσουμε να οργανώσουμε ε, συζητήσεις δημοσιονομικών δημοσιονομικού προσανατολισμού την ίδια εποχή την πρώτη ημέρα να συζητάμε όλοι μαζί και στη συνέχεια ο καθένας στα πλαίσια του Εθνικού του Κοινοβουλίου. Την πρώτη ημέρα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα γίνει μία συζήτηση μεταξύ των 28 ε, κοινοβουλίων, 27 εθνικά συν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καθένας άμενε στη χώρα του, αλλά έχουμε τη δυνατότητα της βίντεο μετάδοσης και θα συζητούσαμε από κοινού για τις ε, δημοσιονομικές ε, αρχές, διότι η οργάνωση αυτής της συζητήσεως θα είχε διάφορα ουσιαστικά προσόντα. Καταρχήν θα μας υποχρεώνε να ξεκινάμε από τις ίδιες οικονομικές υποθέσεις και προβλέψεις όσον αφορά το ποσοστό ανάπτυξης, την τιμή του ευρώ, την τιμή ε, του βαρελιού πετρελαίου, των επιτοκίων ενώ αυτή τη στιγμή σε κάθε χώρα μας ξεκινάει ο καθένας με ε, προκαταρκτικές διαφορετικές ε, υποθέσεις που βολεύουν τον εκάστοτε Υπουργό Προϋπολογισμού. Θα είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και δεσμευμένοι να ξεκινάμε από την ίδια βάση. Δεύτερον, αν γίνει από κοινού αυτή η κίνηση, ο καθένας θα υποχρεούτο να πει ότι ορίστε πως θεωρώ ότι η δημοσιονομική μου πολιτική πρέπει να υπακούει στις ε, ε, ευρωπαϊκές αρχές. Ε, παραδείγματος χάρη στο σύμφωνο σταθερότητος και αναπτύξεως το οποίο θα χρειαστεί να ενημερωθεί για να λάβει υπόψη την οικονομική κρίση αλλά ορισμένα δεδομένα θα παραμείνουν και επίσης θα υποχρεωθούμε ο καθένας από μας να εκφράσει πόσο στον προϋπολογισμό του θα διατηρήσει τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών που προετοιμάζουν το μέλλον ε, της κατάρτισης, ε, της ανάπτυξης, δηλαδή θέματα από των οποίων έχουμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά που θα τελεσφορήσουν μόνο αν αφομοιωθούν σε, όλα τα σε όλους τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα πρέπει κατόπιν συζητήσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να απομειωθούν στο εθνικό, από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινάμε με μία από κοινού συζήτηση και κατά αυτόν τον τρόπο θα έπεφταν τα στεγανά τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ευρώπη. Έχουμε καταργήσει όλα τα σύνορα, όλους τους ελέγχους. Υπάρχει ακόμη όμως ε, ένα εμπόδιο που διατηρεί τη δημοσιονομική συζήτηση σε εθνικό επίπεδο ακόμη και αν οι κατευθύνσεις διατυπώνονται από κοινού από τις 27 κυβερνήσεις στις Βρυξέλλες. Εάν λοιπόν προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε μία τέτοια δυνατότητα χωρίς ε, καμία περαιτέρω νομική υποχρέωση θα πρόκειται για μία ανταλλαγή απόψεων περίπου όπως σήμερα. Και πιστεύω ότι μία τόσο απλή διαδικασία θα έχει το προσόν να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προσπαθίας ε, συγκρίσεως και συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών εξασφαλίζοντας ότι θα εμπλέκονται τα εθνικά κοινοβούλια απαρχής και στη συνέχεια θα δούμε ότι κάθε κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό ε, ε, Συμβούλιο θα καταρτίζουν τα συνολικά, τους συνολικούς προϋπολογισμούς. Αυτή είναι όμως μία απρή πρόταση την οποία θέλω να υποβάλω. Έχουμε βέβαια και άλλους εγγεγραμμένους Υπάρχει μια Ιταλική αντιπροσωπεία σημαντική, την οποία χαιρετίζω επίσης, μεταξύ των οποίων είναι ο κύριος Καραβάλια της Ιταλικής Γερουσίας, ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Εκπροσωπώ την Ιταλική Γερουσία και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μα δίνετε σε αυτή, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι πιθανέ συνέργειε ανάμεσα στον ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό και στου Εθνικού προπολογισμού και στη συνέχεια ε, να σα μιλήσω για τη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή Προπολογισμού σε σχέση με τον, ε, της Γερουσίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, συμφωνούμε με τον κύριο Λαμασούρ με βάση τη μελέτη που έγινε πραγματικά, ε, ενώ είναι γίγαντα από νομική άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι νάνο όσον αφορά τον προπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπάρξουν ισχυρέ συνέργειε ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και στου Εθνικού, ακριβώ γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Με εξαίρεση τα διορθωτικά ταμεία, η μελέτη δεν ε, εντόπισε σημαντικέ μορφέ ε, συντονισμού ανάμεσα στην, στη, στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στου εθνικού προπολογισμού, που παραμένουν δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Αυτό φαίνεται ε, και μέσα από ορισμένε ε, ε, συγκεκριμένα παραδείγματα όπου φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε εθνικό επίπεδο δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την προσθέμενη αξία σε, ευρωπαϊκό, επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι διαποτισμένο από, από ένα πολιετή προγραμματισμό που είναι ιδιαίτερα άκαμπτο. Ενώ οι εθνικοί προπολογισμοί στηρίζονται σε εθνικό εθνικό προγραμματισμό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τον προγραμματισμό. Τώρα, ποιε είναι οι πιθανέ συνέργειε ανάμεσα στου εθνικού προπολογισμού και στον ε, ε, ευρωπαϊκό. Η μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού είναι ε, ασθενή, γιατί ακριβώ δεν είναι ιδιαίτερα δεσμευτική. Και οι βασικέ κατευθυντήριε γραμμέ οικονομική πολιτική. Ενδιαφέρουσα αυτή η πρότασή σα για μια προκατακτική συζήτηση. Ε, και ε, πραγματικά ε, να έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία προ την κατεύθυνση αυτή θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Όσον, κοίταξε, αυτή τη στιγμή θέλουμε να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο και από τι ενέργειε. λαμβάνοντα υπόψη και την προσπάθεια που καταβάλουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. η έλλειψη πόρων μπορεί να, ορίσει, να, να οδηγήσει τα Υπουργεία στο να κατα, καταρτήσουν λεπτομερεί καταλόγου προτεραιοτήτων και να δούμε πώ μπορεί να υπάρξει η, η σχέση με με, το, με, την, με τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή όσο δίνεται τι πιθανέ συνέργειε. Εξάλλου, λαμβάνοντα υπόψη ε, ότι εμεί είμαστε καθαρό συνεισφέρον, ε, θα μπορούσαμε να ε, αντλήσουμε ιδιαίτερη ε, προστέμενη αξία από τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Τέλος, ε, σας λέω ότι ε, θα μπορούσαμε ε, να εντοπίσουμε συγκεκριμένα το που υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα σε εθνικές πολιτικές και στις πολιτικές που υλοποιούνται με βάση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς προτείνουμε να γίνει αυτό με, αναλύοντας το Ιταλικό παράδειγμα. Πρέπει να σας πω ότι σε επίπεδο γερουσίας γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση με, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από αυτά τα χρόνια εμπειρία ε, τη Νομισματική Ένωση, φαίνεται ότι αυξήθηκαν οι ανισορροπίε σε οικονομικό επίπεδο ανάμεσα ε, στα κράτη-μέλη. Η, η ευκταία σύγκληση δεν επετεύχθη. Εξακολουθούν να υπάρχουν τομεί όπου συσσωρεύονται τα ελλείμματα ε, στα, εμπορικά ισοζύγια και στον τομέα τη παραγωγικότητας παραγωγικότητα. Ενώ ε, άλλε χώρε έχουν εμπορικά πλεονάσματα. Αυτή η διαδικασία λοιπόν τη σύγκληση πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Διαφορετικά ε, θα, θα τεθεί σε κίνδυνο η ίδια ύπαρξη του ευρώ. Η μέγιστη πιθανή σύγκληση αποτελεί λοιπόν ε, μια προτεραιότητα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τα προσεχή χρόνια. Η αύξηση των πιστώσεων για την ανταγωνιστικότητα και για την συνοχή είναι κάτι το πολύ σημαντικό γιατί θα βοηθήσει ε, προ την κατεύθυνση αυτή. Τέλο, κατά τη συζήτηση για την ε, έγκριση του πολιετού δανείου προ την Ελλάδα, ε, είδαμε το πώ αυτό αποτελεί ένα, ένα, ένα θεσμικό στοιχείο για την Ευρώπη. Δηλαδή, πολλά κράτη-μέλη πρέπει να πούμε, μάλλον θα πρέπει να πούμε μου ότι η σωτηρία ε, της, ε, της Ελλάδας είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, παρά το γεγονός ότι προέρχονται και κονδύλια ε, από, ε, από αλλού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό, όπως τον βλέπουμε σήμερα, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής αλλαγής στο προσεχές μέλλον. Καλό λοιπόν την Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω άλλωστε ελέγχθηκε πριν από λίγο, να ε, αφιερώσει μία σύνοδο εργασία ε, για τη μελέτη αυτή τη πτυχή ε, και να συμμετάσχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Μιλώ για αυτή τη νέα προοπτική που θα πρέπει να λάβει ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε για τη συμβολή σα, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καρέ ο οποίο εκπροσωπεί την ε, Γαλλική Συνέλευση. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ για την ε, ε, διοργάνωση αυτή τη συνεδρία που είναι πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Το είπατε κι εσεί ότι είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική αυτή η στιγμή όπου αντιμετωπίζουμε σοβαρές, σοβαρή κρίση και ο καθένα καταλαβαίνει ότι πρέπει να σταθεί στο ύψο των αποφάσεων που θα ληφθούν. Ταυτόχρονα να σας πω ότι ε, κάνατε συγκεκριμένε προτάσει, πράγμα που δεν, είναι, που δεν γίνεται πάντα. Ε, μέσω λοιπόν του εγγράφου σα, το οποίο σα λέω ότι και σε προσωπικό επίπεδο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, θα μπορούσαμε ε, να αντιδράσουμε όλοι μαζί. Τώρα, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά του στόχου. Συμφωνώ με την άποψή σα. Πιστεύω ότι πράγματι εδώ έχουμε δύο βασικέ απαιτήσει. Και κάθε μία από τι ευρωπαϊκέ χώρε θα πρέπει να τι αντιμετωπίσει. Η πρώτη είναι προφανώ να, η, εξη, ε, εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών είναι σαφώς ε, επιτακτική ανάγκη και δεύτερον να διατηρηθεί και η ανάπτυξη, μην το ξεχνάμε, γιατί Λαμβάνοντας υπόψη τις κυρώσεις που ε, επιβάλλουν οι αγορές στις χώρες, εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Ε, βεβαίως ε, υπάρχει το θέμα των ελλημάτων, αλλά από την άλλη είναι μικρή ανάπτυξη ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η συμφιλίωση λοιπόν αυτών των δύο στόχων είναι δύσκολο, γιατί μέχρι στιγμή και αυτό ελέγχθη άλλωστε, αυτό δεν κατέστη δυνατό με ικανοποιητικό τρόπο κυρίω όσον αφορά τη σύγκληση των οικονομιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία δεν επετεύχθη. Άρα πράγματι θα πρέπει να εφεύρουμε νέα εργαλεία. Και να σα πω το εξή, και εδώ συμφωνώ και με την ανάλυση σας βεβαίως, ε, προφανώς ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ισχυρή δυνατότητα παρέμβαση τη Ευρώπη, εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο σα έλεγα, την ε, ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ορισμένε προτάσει. Ε, ε, να σα πω κάτι το οποίο είναι προσωπική μου άποψη. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε να υπάρξει και ίδια διαφορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον προπολογισμό. Δεύτερον, όσον αφορά τον συντονισμό. Και εδώ είναι επιτακτική ανάγκη, σαφώ. Ε, το βλέπουμε. Η απουσία δημοσιονομικού συντονισμού ε, δεν μπορεί να διατηρηθεί πλέον. Άρα θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο προ την κατεύθυνση αυτού του συγκεκριμένου συντονισμού, λαμβάνοντα υπόψη και τελώντα αντιτάγματα διδάγματα ε, ε τη εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Λαμβάνοντα υπόψη δηλαδή ότι αυτό ο συντονισμό μέχρι στιγμή δεν κατέστη λειτουργικό. Έχουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι δεν έγινε πάντα κατανοητή στο βαθμό που θα έπρεπε. Ίσως γιατί δεν ε, εξηγήθηκε σωστά. Πάντως σε προσωπική βάση σας λέω ότι δεν με εκπλήττει αυτή η πρόταση. Αλλά είναι αλήθεια ότι στη χώρα μου ε, δεν έτυχε καλή υποδοχή, ε, γιατί ορισμένοι θεώρησαν ότι αποτελεί πλήγμα στην εθνική κυριαρχία. Πάντω σα λέω ότι είναι σαφέ ότι θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο ε, όσον αφορά αυτό το συντονισμό και νομίζω και εδώ είναι ενδιαφέρουσα η πρότασή σα. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, και ανεξάρτητα από το μέσο που θα επιλέξουμε, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να εμπλέκονται πολύ περισσότερο. Αυτό για μένα είναι απαραίτητη προπόθεση. Και από την άποψη αυτή, η πρότασή σα, η ιδέα αυτή αυτής της ετήσιας διακοινοβουλευτικής συνδιάσκεψης μου φαίνεται πολύ σωστή. Διότι θα επιτρέψει την αδιαφυσβήτη υπέρβαση ορισμένων δισταγμών και επιφυλάξεων, Όπω αυτέ που εκφράστηκαν στη χώρα μου απέναντι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή επιτροπή. Είναι καλό αυτό ο δρόμο λοιπόν, είναι σωστή η πρόταση και σα λέω ότι ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου τη Γαλλία, παρόλο που δεν έχω την επίσημα την αρμοδιότητα και την αξιοδότηση να μιλήσω για λογαριασμό του, πάντω σα λέω ότι σίγουρα ε, θα αντιδράσουν θετικά τα μέλη του Κοινοβουλίου μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Μια και εδώ ακόμα οι Γερμανοί φίλοι. Σα κάνουμε ρησία σας. μίλησαν εκπρόσωποι τριών κοινοβουλίων Γερμανίας, Ιταλίας και, και Γαλλίας των τριών δηλαδή μεγαλύτερων οικονομιών της ζώνης του ευρώ και της υπηρετικής Ευρώπης. Πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν πολύ διαφορετικές συνθήκες προς την ανταγωνιστικότητά τους. Το εξωτερικό τους ισοζύγιο, και τα δημοσιονομικά τους. Πλην όμως και οι τρεις χώρες πάσχουν από μια κοινή νόσο ασθενική ανάπτυξη. Και οι τρεις αυτές χώρες, οι πιο σημαντικές οικονομίες της όρης του ευρώ, οι χώρες εκείνες οι οποίες θα πρέπει να παρασύρουν προς τα μπρος τις άλλες οικονομίες, έχουν δυστυχώς ραχητική ανάπτυξη τα 7 πρώτα έτη του 21ου αιώνα, πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια των πρώτων 7 ετών και πριν από την εκδήλωση της κρίσης, το είπα και νωρίτερα και το ξαναλέω, τα, τα 7 αυτά πρώτα έτη ήταν τα πιο... Ε, τα κράτη με τις μεγαλύτερες για ολόκληρο τον κόσμο. 3, 4, 5, 6, 7% ανάπτυξη είχαν τα κράτη της Ασίας, 5, 6% της Λατινικής Αμερικής οι Ηνωμένες Πολιτείες 3%, η Αφρική 4-5%. Ακόμα και φέτος μετά την κρίση η Αφρική έχει 5% ανάπτυξη. Τα κράτη αυτά όμως τα τρία τα ευρωπαϊκά είχαν 1% μέσο όρο ανάπτυξης για 7 χρόνια, τα 7 χρόνια πριν από την εκδήλωση της κρίσης. Αυτή είναι η κοινή νόσος που καλούμαστε να θεραπεύσουμε. Παρ' όλα αυτά είχαν και διαφορετικές στρατηγικές τα τρία αυτά κράτη. Καταλαβαίνω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Γερμανοί φίλοι Φερρυπίν όταν συγκρινόμενη η Γερμανία με τη Γαλλία για την ίδια περίοδο και βλέπουμε ότι οι Γάλλοι αποφάσισαν, οι Γερμανοί αποφάσισαν να κάνουν περισσότερες προσπάθειες την περίοδο που οι, Γερμαν, οι Γάλλοι αποφάσισαν να σταματήσουν να κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες. Επτά χρόνια μετά η Γερμανία μπορεί να είναι η πιο ανταγωνιστική χώρα του κόσμου, η πρώτη χώρα εξαγωγών μας με την ε, Κίνα, αλλά ο εθνικός της πλούτος, το ΑΕΠ της, έχει πολύ βραδία ανάπτυξη. Δηλαδή δεν έχουν μπορέσει να διαφοροποιηθούν από τους Γάλλους, δηλαδή δεν έχουν μπορέσει να μειώσουν την ενεργεία τους, δεν έχουν μπορέσει να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και το δυναμικό ανάπτυξη, ακόμη και μετά το τέλος της κρίσης με βάση προβλέψεις των ε, οικονομολόγων θα μείνει πάλι στο 1%. Η Γαλλία χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες, με απώλεια ανταγωνιστικότητας, φτάνει και πάλι σε πολύ απογοητευτικά ποσοστά ανάπτυξης, χωρίς να τολμώ να κρίνω τα ποσοστά της Ιταλίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι και για τα ίδια αυτά 7 έτη η Ιταλία σημειώνει μηδενική ανάπτυξη, ενώ ο κόσμος καλπάζει, η παγκόσμια οικονομία καλπάζει. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, διότι όσο δεν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 2,5-3% που να διατηρούνται για αρκετά χρόνια, δεν μπορούμε να μιλούμε για χρηματοδότηση των συστημάτων συνταξιοδότησης, για ανάκαμψη των δημοσιονομικών, για ανταγωνιστικότητα στο εγγύης μέλλον. Και ως εκ τούτου πρέπει να συζητήσουμε με σοβαρότητα, διότι υπάρχει πρόβλημα, θα έλεγα, επιστημονικού χαρακτήρα. Ποια είναι η καλή οικονομική πολιτική, το καλό policy mix, όπω το λέγαμε τώρα, χρηματοδότηση των επενδύσεων για το μέλλον και δημοσιονομική πολιτική και βέβαια και νομισματική πολιτική μαζί. Και επίση, πολιτική ισορροπία ή καλύτερα πολιτική εξίσωση, που θα πρέπει να διατυπώσουμε έτσι ώστε να πείσουμε και τις ε, κοινέ μας γνώμες για τις επιλογές που θα κάνουμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Εμπνέομενοι ασφαλώς και από τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Μένωσης που είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τίμες. Αυτά ως προσωπική παρατήρηση. Αφού ακούσαμε τρεις συνάδελφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ας ακούσουμε και τον Σαλβαδόρ Γαρίγα, ε, επιφανή συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ε, υπηρετική Ευρώπης, την Ισπανία. Παρακαλώ. Ε, μου ε, αναφέρετε μεγάλη ευθύνη κύριε Πρόεδρε. Πάντως ε, θέλω να τοποθετηθώ εξ ονόματος ε, των ε, μελών του Κοινοβουλίου μας που δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα ακριβώς λόγω ε, δημοσιονομικών περικοπών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό το θέμα της συζήτησης σήμερα και θα πρέπει να πάρουμε το λόγο για να εκφράσουμε μια κοινή θέση. Εκφράζω λοιπόν κοινή θέση εκ μέρους των συναδέλφων του κοινοβουλία μας. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπατε κύριε Λαμασούρ για τη σημερινή ημερίδα συζητήσεων και, και για την ημερίδα που θα διοργανώσουμε για να μιλήσουμε ε, για τους ε, που, που οργανώσαμε μάλλον για να μιλήσουμε για τους ε, προσανατολισμούς ε, του ε, προπολογισμού. Και είναι σημαντική αυτή η συνάντηση για να καταλάβουν όλοι μέχρι ποιο σημείο υφίσταται αυτή η ισχυρή αντίφαση ανάμεσα στους κοινοτικού στόχου και στα κοινοτικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την επίτευξη των στόχων αυτών που από την άλλη μεριά συμφωνήθηκαν στα διάφορα ευρωπαϊκά συμβούλια. Ε, στόχοι των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που στη συνέχεια μετά από τα ευρωπαϊκά αυτά συμβούλια οι πρωθυπουργοί των κρατών μελών έρχονται στα εθνικά κοινοβούλια και εξηγούν τους στόχους αυτούς. Ε, εξηγούν λοιπόν ε, στα μέλη του Κοινοβουλίου του στόχου οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, αλλά ποτέ δεν μιλούν για τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σα το λέω γιατί εγώ υπήρξα μέλο του Εθνικού Κοινοβουλίου και όπω είπε και ο συνάδελφο από την Ιταλία, πολλέ φορέ ε, ε ω εθνικοί βουλευτέ ε, αναρωτιόμασταν ε, για το πόσο. δεν δε δεν, ασχολιόμασταν μάλλον για το τι θα, συνεπα, τι θα σήμεναν αυτές οι δεσμεύσεις ε, οι ευρωπαϊκές, αλλά πόσο θα μας κόστιζαν. Και τέλο, αυτή η κοινή συζήτηση ανάμεσα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια ε, αποτελεί τη βάση έτσι ώστε να εξηγηθούν οι προτεραιότητε, ε, να εξηγήσουμε δηλαδή τι προτεραιότητε και να εξηγήσουμε και ότι πολλές φορές εμεί ερχόμαστε σε σύγκρουση με το Συμβούλιο γιατί λοιπόν μερικές φορές για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του προπολογισμού ε, μιλάμε τελικά ε, για το μέσο ευοληξίας, εκεί φτάνουμε και ε, αγωνιζόμαστε σκληρά στο Συμβούλιο για να πετύχουμε αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ε, για το μέσο ευελιξία, γιατί, χρειαζόμαστε γιατί χρειαζόμαστε ταυτόχρονα περισσότερα χρήματα για το Ταμείο ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, για το μέσο αλληλεγγύη κτλ. Αλλά πέραν όλων αυτών, που έχουν να κάνουν με την ε, ε, τεχνική, τη δημοσιονομική, την καθημερινή. Θέλουμε κυρίω τα εθνικά κοινοβούλια να κατανοήσουν και να μα υποστηρίξουν, έτσι. Γιατί σε τελευταία ανάλυση τα μέσα μα, όπω αναφέρει και το έγγραφο Λαμασούρ, ε, τελικά τι είναι. Ε, είναι ε, αν θέλετε, ε, ε μια, ε, ε, αυτά που ζητάμε είναι παραχωρήσει από του εθνικού προπολογισμού που τους συμφωνούν οι εθνικοί βουλευτέ και όχι οι, Ευρωπαίοι. Κυρίω όμω θέλω να κατανοήσουν τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια το ε, πώ γίνεται η εξέταση του προπολογισμού και αυτό το θέμα και το γιατί αυτό το θέμα ε, δημιουργεί τρομερά, τρομερά προβλήματα και συγκρούσει. Αλλά όλα αυτά έχουν νόημα και θέλουμε να το κατανοήσουν. Μόνο να ακολουθήσουμε την πρόταση Λαμασούρ. Δηλαδή να, να υπάρχει εκ των προτέρων μια γνήσια συζήτηση έτσι ώστε να κατανοούμε όλοι ε, πώ οι εθνικοί προπολογισμοί ε, είναι συμβατοί με, τις βασικές, ε, του βασικού προσανατολισμού που αποφασίζονται στι Βρυξέλλε. Αν δεν υπάρχει συνεχή ροή πληροφοριών και επικοινωνία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε τελευταία ανάλυση οδηγούμεθα σε μια κατάσταση έλλειψη εμπιστοσύνη, αντίδραση, αντίσταση. Ε, ε, ο καθένα οχυρώνεται γύρω από τι δικέ του αρμοδιότητε και δεν μπορεί να υπάρχει συντονισμό των προπολογισμών. Γι' αυτό πιστεύω και ε, εκφράζω και την ιδέα των, των Ισπανών εκπροσώπων ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει σήμερα ομοφωνία γύρω από την ιδέα Λαμασούρ όλων των συμμετεχόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σαλβαδόρ έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών και Δημοσίων Δαπανών της Δίαιτας της Πολωνίας, στον οποίο δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την συνεδρίαση αυτή και την ευκαιρία που μας προσφέρεται τα προβλήματα του συντονισμού των προπολογισμών και της αποτροπής της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι από τα πιο σημαντικά που έχουμε. Και με ικανοποίηση βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στρατευτεί στο σκοπό αυτό. Έχουμε και εμείς στην Πολωνία ε, συζητήσει τα θέματα αυτά Φαίνεται ότι έχουμε μπορέσει να διέλθουμε την κρίση με λιγότερα προβλήματα από ότι, τα άλλα κράτη-μέλη, από ότι κάποια άλλα κράτη-μέλη. Μεν, πλην όπω γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι τα προβλήματα είναι κοινά και μα επηρεάζουν όλου και μπορεί να επηρεάσουν και την Πολωνία στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον να ακούμε όλε τι ιδέε που ενδεχομένω ακουστούν για τον τρόπο αποτροπή των προβλημάτων, αντιμετώπιση του επίση. Αλλά πάνω απ' όλα η πρόληψη μα ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αποτρέψουμε, να προλάβουμε την οικονομική κρίση και βέβαια τα ζητήματα της δημοσιονομικής πειθαρχία. Είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Βλέπουμε ότι κράτη που δεν έχουν δημοσιονομική πειθαρχία μπορεί να υποστούν κυρώσεις είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, αλλά εάν πρόκειται να επιβληθούν τέτοιου είδους κυρώσεις, απαιτείται αυτές να είναι και δίκαιες. Αυτό το λέω διότι φάνηκε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εννοεί ότι τέτοιου είδους ε, κυρώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και πάυση ε, πληρωμών από τα ταμεία συνοχής, από τα ταμεία συνοχής, περιοριστικά ταμεία, πράγμα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο διότι αυτά, αυτά ε, τέτοιου είδους κυρώσεις θα απέβαιναν εις βάρος και θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στα πιο φτωχά κράτη-μέλη. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν είμαστε κατά των κυρώσεων, απλώς επιμένουμε ότι αυτές θα πρέπει να αφορούν όλα τα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως των ε, κονδυλίων ή των ταμείων των οποίων επωφελούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η στρατηγική του 2020 επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως τρόπος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερα η έρευνα και η ανάπτυξη ασφαλώς θα διαδραματίσουν εδώ πολύ ε, σημαντικό ρόλο, πρέπει να αποτελέσουν για το μέλλον προτεραιότητες όλων μας και βέβαια ναι, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε και να δράσουμε, υπενθυμίζοντα όμως ταυτόχρονα ότι μακροπρόθεσμα και στην πράξη αυτό ίσως να έχει σαν συνέπεια πως κάποια οι περιφέρειες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτυχθούν πιο γρήγορα από κάποιες άλλες που θα μείνουν πίσω. Και έτσι Καλό θα ήταν πιστεύω να εξετάζουμε όχι μόνο που υπάρχουν τα σημαντικά κέντρα, τα ερευνητικά, τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά να ε, έχουμε πάντα υπόψη και τη γεωγραφική κατανομή, έτσι ώστε η έρευνα και η ανάπτυξη να αναπτύσσονται κατά τρόπο ομοιόμορφο στις διάφορες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισμός των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο όπως άλλωστε μας επεσήμανε και ο πρόεδρος τομείς που θα μπορούσαν ε, να τύχουν συντονισμού στον, ε, στους προϋπολογισμούς μας ε, είναι Φερρυπίν όσον αφορά την Πολωνία, αλλά και άλλες χώρες ασφαλώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφορά αυτό, το ζήτημα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Εμείς πληττόμεθα από τακτικές πλημμύρες, Φερρυπίν. Και έτσι ίσως θα μπορούσαμε από τα δημόσια μας ε, προγράμματα ε, να συντονίσουμε τις επενδυτικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, για την υπερσυνοριακή ή ε, καθαρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις έτσι ώστε προσπάθειες που κάνει μια χώρα να μην επαναλαμβάνονται από κάποια άλλη χώρα. Και πάλι στόχος μας εδώ είναι η πιο αποτελεσματική κατά το δυνατόν δράση. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στον τομέα των υποδομών των μεταφορών ή στην ασφάλεια σε προμήθεια ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δημοσιονομικός λοιπόν συντονισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάντα όμως και με γνώμονα την αρχή της επικουρικότητας. που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αντικαταστήσει στις δράσεις αυτές τις εθνικές αρχές. Μόνο συμπληρωματικό ρόλο, ρόλο αρρωγής μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ρόλο που θα ενισχύσει τις ε, οικονομίες, τους προϋπολογισμούς μας και έτσι στο μέλλον ε, να μας επιτρέψει να συζητούμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα συντονισμού του ευρωπαϊκού με τους εθνικούς προπολογισμούς. Ο κύριος Λαμασούρ. Νομίζω ότι όλοι εντυπωσιαστήκαμε από τις οικονομικές επιδόσεις της Πολωνίας το 2009 που ήταν η μόνη ευρωπαϊκή οικονομία που διετήρησε μία θετική πορεία και ελπίζουμε ότι όλοι θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά σας και θα τα καταφέρουμε κάπως καλύτερα εφέτος. Μία άλλη χώρα που έχει ένα πρότυπο αναπτύξεως που αντιμετωπίζει δυσκολίες είναι η Σουηδία και δίνω τον εκπρόσωπο στον Γκόραν Φέρν, ο, ο οποίος είναι ε, σοσιαλιστής ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ. Δεν είμαι αντιπροσωπευτικός για τη Σουηδία γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική μου ομάδα είναι στην αντιπολίτευση στη Σουηδία. Ελπίζω όχι για πολύ ακόμη αλλά τέλος πάντων. Πρόεδρε, ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και νομίζω ότι καλό θα ήταν τώρα να ασχοληθούμε με την όθηση η οποία έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή ε, δεν πρέπει να σπαταλήσουμε μια καλή κρίση η οποία ε, βοηθάει και αυτό θα πρέπει να, να ληφθεί υπόψη. Βέβαια χρειάζεται να συζητήσουμε την κρίση κίνηση αυτή. Υπάρχουν ορισμένες πολιτικές είδατε ότι την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο νέος Υπουργός Οικονομικών στο Ηνωμένο Βασίλειο έφεσε βέτο για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η αύξηση του προϋπολογισμού, αυξημένη φορολογία είναι θέματα που δεν μπορούν να προχωρήσουν τώρα. Η συζήτηση ε, ε, πρέπει να προχωρήσει σε εφόλης της και και εδώ όπως και στα κράτη-μέλη. Και η σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ή άλλως καταρτίζει ένα έγγραφο για την δημοσιονομική μεταρρύθμιση ε, πράγμα το οποίο έχει κινητοποιήσει την εθνική μας αντιπροσωπεία διότι ε, σε εποχή κρίσεως χρειάζεται να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη, για τις θέσεις εργασίας, για τις δράσεις σταθερότητος, χρειαζόμαστε συνεργασία για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η κοινωνία όπως ε, ε, είπατε λόγω των κλιματολογικών αλλαγών, ε, λόγω των διαφόρων τάσεων που διαγράφονται. Οπότε παρόλες τις τους δημοσιονομικούς περιορισμούς έχουμε όλο και περισσότερες ενέργειες αλλά όλο και λιγότερους σπόρους. Αν δείτε λοιπόν την κλιματική πολιτική, την καταπολέμηση της εγκληματικότητος, όλα αυτά είναι δαπανηρά εγχειρήματα και ασύμβατα. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι που λέγουν εφόσον έχουμε νέες προτεραιότητες θα καταργήσουμε τις παλιές. Αλλά εάν περιορίσουμε παραδείγματος χάνει την κοινή γεωργική πολιτική βλέπουμε ότι ορισμένοι αρνούνται ή αν μειώσουμε ε, την πολιτική συνοχή, διότι πλουταίνουν οι χώρες δεν χρειαζόμαστε τόσο την πολιτική συνοχής απ' την άλλη πλευρά διευρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με πιο φτωχά μέλη οπότε ούτε αυτό είναι λύση άρα τι πρέπει να κάνουμε <clears throat> επειδή ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες ε, πρέπει να πω ότι υιοθετώ τις απόψεις του Προέδρου μας και πρέπει νομίζω να κάνουμε ορισμένα πράγματα να εστιαστούμε σε μια βελτιωμένη ποιότητα των δαπανών και να μπορέσουμε να αποκομίσουμε περισσότερα ξεκινώντας από λιγότερα ε, καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν διότι ε, ε, πρέπει να είναι συμπληρωματικός ο εθνικός προϋπολογισμός με τον κοινοτικό θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη προστιθέμενη αξία από, την, ε, από συνοριακές ε, ε, επενδύσεις, από συνεργασίες. Ας εστιαστούμε σε οικονομίες μέσω του ευρωπαϊκού συντονισμού, διότι ουσιαστικά θα έπρεπε να μειώσουμε το κόστος της εθνικής διοικήσεως με την εμπλοκή της ευρωπαϊκής διοικήσεως, αλλά δεν είναι προφανές και θα πρέπει να βρεθούν ε, εθνικές οικονομίες εφόσον χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκές δυνατότητες. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να προωθήσουμε και νέες μεθόδους για την αποκόμιση ε, εσόδων κατόπιν συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Ε, εμείς ε, νομίζω πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα της ανεξάρτητης φορολογικής αρμοδιότητας σε εθνικό επίπεδο. Αυτό δεν λειτουργεί. Ναι, ε, ε, πρέπει να σεβόμαστε τις εθνικές φορολογικές ιδιομορφίες, αλλά είναι και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Διότι βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να πληρώσουν για τις νέες ενέργειες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά ευχαρίστως να πληρώσουν για τον ειδικό μηχανισμό για τις κλιματολογικές αλλογές ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια για διάφορους τομείς σε όλα αυτά υπάρχει λιγότερη διαφάνεια υπάρχει λιγότερη δυνατότητα καταρτήσεως προ μίας λίστας προτεραιοτήτων βάσει ορθολογιστικής σκέψης και υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Ίσως λοιπόν Δίκιο έχει ο Πρόεδρος ότι πρέπει να συναντιόμαστε πιο τακτικά και πιο οργανωμένα μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σε σχέση με αυτό που είπε ο Φέρμ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, απέναντι σε αυτή την επίγουσα κατάσταση, οι κυβερνήσεις μας πρέπει να λάβουν ορισμένε αποφάσεις. με τους οποίους μπορεί να συμφωνούμε ορισμένοι, αλλά κάτω από ε, προϋποθέσεις και συνθήκες που διαφεύγουν του παραμικρού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και βεβαίως δεν μπορούμε επομένως να εγκρίνουμε τη διαδικασία, μπορούμε να συμφωνούμε επί της ουσίας, αλλά ως ε, κοινοβουλευτικοί, ως, ε, ως εκλεγμένοι από τους πολίτες για την ε, ε, για να σεβόμαστε και τα εθνικά συντάγματα αλλά και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση. Παράδειγμα. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα και από πλευρά δαπανών και από πλευρά εσόδων. Όσον αφορά τι δαπάνε. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιανουαρίου αναφερόμενοι στην πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια στην αποτυχία της συνδιάσκεψης Κοπενχάγης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει, να εφαρμόσει μία πρόταση που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την Κοπεχάγη στην περίπτωση που θα ε, πετύχαινε η Κοπενχάγη και που συνιστάται στο να βοηθήσουμε τι αναψώμενε χώρε να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή με οικονομική δηλαδή βοήθεια ευρωπαϊκή τη τάξη των 2,5 δι ευρώ. 2,5 δις ευρώ. Άρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε και το μάθαμε μέσα από μια ανακοίνωση τύπου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εν τη σοφία του αποφάσισε να δώσει το 2010, από το 2010 έτσι, 2,5 δις ευρώ στις αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Και αυτό το ποσό θα ανανεωθεί το 2011-2012 και στη συνέχεια θα προσαυξηθεί. Θα είναι το ίδιο λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια και δεν θα αυξηθεί. Όταν τα ακούσαμε, κοιτάξτε, ε, καταλαβαίνετε τα συναισθήματά μα. Ε, και ρωτήσαμε τι γίνεται και μα είπαν, μα δεν σα αφορά, δεν είναι χρήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα, θα προέρχονται τα χρήματα αυτά από του εθνικού ε, προπολογισμού. Συμφωνήσαμε εμεί οι κυβερνήσει να μοιραστούμε το ποσό αυτό σύμφωνα με μια κλίδα κατανομή που τη διαπραγματευτήκαμε μεταξύ μα μια κλίδα κατανομή που σε γενικέ γραμμέ αντιστοιχούσε στο ΑΕΠ καθένα, κρατών μελών. Πάντως το καθένα από τα κράτη-μέλη πάντως το διαπραγματεύτηκαν από κοινού οι κυβερνήσεις. Να λοιπόν ένα παράδειγμα απόφαση που έλαβαν οι, αρχι, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων στι Βρυξέλλες και που διέφυγε τελείω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Και φοβάμαι και ότι διέφυγε και του μεγαλύτερου μέρου των εθνικών κοινοβουλίων. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, κάθε εθνικό κοινοβούλιο εξετάζει και εγκρίνει το εθνικό μερίδιο που αφορά αυτή τη συνολική πολιτική. Αλλά για να κρίνει κανεί τι επιπτώσει αυτή τη συνολική πολιτική, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να κρίνει το τι θα δώσει η Σλοβενία, αν θέλετε. Το, το τη Σλοβενία θα δώσει η Σλοβενία ή τη Γαλλία θα δώσει η Γαλλία. Αλλά συνολικά δηλαδή να αξιολογήσουμε την πολιτική αυτή. Άρα λοιπόν να βλέπετε ότι έχουμε να κάνουμε μια σημαντική πολιτική η οποία διέφυγε πραγματικά του κοινοβουλευτικού ελέγχου τόσο στις Βρυξέλλες όσο και σε εθνικό, και σε επίπεδο. Να δώσω και άλλο παράδειγμα. Νομίζω ότι 21-22 χώρες από τις 27 στείλαμε στρατιωτική βοήθεια στο Αφγανιστάν. Κανένα από τα κοινοβούλια μας δεν μπορεί να ασκήσει πολιτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της πολιτικής αυτής. Δηλαδή ο καθένα βλέπει τα πράγματα με τη σκοπιά τη δική του ερωτική ποσότητα. Αυτό από μεριά δαπανών. Εσόδων τώρα. Από μεριά εσόδων. Μάθαμε, νομίζω όλοι με ικανοποίηση και με ανακούφιση, ότι στι 9 Μαου 2010 οι κυβερνήσει μα συμφώνησαν στο σχέδιο οικονομικής διάσωσης με αυτό το οικονομικό απόθεμα με τη μορφή ε, ε, δυνατότητας ε, δανείου 50 δις ευρώ. Συγγνώμη, 550 δις ευρώ. Λοιπόν, όσον αφορά τα χρήματα αυτά, ε, ικανότητα, έχουμε και την ικανότητα δανειοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μάλιστα. Έχουμε και τα 60 δις που, είναι ικανότητα, που προέρχονται από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα από το Δούνου Διαβάζοντας λοιπόν την, ε, ε, ε, τη συνθήκη βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν είναι δυνατόν δηλαδή θα βρει ε, αυτά τα 60 δις για να βοηθήσει μια, τη χώρα που θα αντιμετωπίζει έκτακτες δυσκολίες. Αυτά τα 60 λοιπόν δις ευρώ δεν θα φανούν πουθενά σε κανένα προπολογισμό. Δεν θα μπορούν να, βρίσκονται, να, να εμφανιστούν, δεν μπορούν να εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό αλλά ούτε και στου εθνικού. Στους εθνικούς θα έχετε το μερίδιο το οποίο θα αφορά τη δική σας ε, τη χώρα. Και η νομική λύση που βρέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την, για την εφαρμογή αυτής της ικανότητας δανειοδότησης και, ε, και δανείου ξεφεύγει από κάθε, κάθε ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι από κοινού. Για να φροντίσουμε έτσι ώστε ο δημοσιονομικός συντονισμός θα επιτρέψει και την εξασφάλιση συμπληρωματικού χαρακτήρα των αποφάσεων που λαμβάνονται και που αφορούν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και, και του εθνικού προπολογισμού, αλλά θα επιτρέψει επί, ταυτόχρονα να υπάρξει ένα πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, δημοκρατικό, με δημόσια συζήτηση, ψηφοφορία, παρουσίαση ε, στην κοινή γνώμη μέσω των, ε, ε, από τα μέσα αυτών των αποφάσεων που έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσει. και που βεβαίω το ξαναλέμε κάτω από την, από την πίεση των εκτάκτων περιστάσεων, έτσι. Ε, ε, εφαρμόζονται σήμερα μέσα από σκοτεινέ διαδικασίε που δεν είναι καθόλου διαφανεί. Και, αυτό πρέπει το, και αυτή η κατάσταση θα πρέπει να, να ομαλοποιηθεί. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντίλιο, ε, εκπρόσωπος από το άλλο σώμα της Ιταλίας, από την Κάτω Βουλή, πάλι από την Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστούμε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον, τον πρόεδρο, τον κύριο Λαμασούρ, για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτηση, την οποία θεωρώ πολύ χρήσιμη. Προσωρινά είμαι πεπισμένος ε, και και αυτό το αναφέρω και σήμερα και επανειλημμένα το έχω πει ότι θα, ε, είμαι πεισμένο λοιπόν για το ότι θα, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό και συνέργεια ανάμεσα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και στου εθνικού προπολογισμού. Ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των ε, πολιτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη. Εδώ ε, αναφέρθηκε και η αρχή της επικουρικότητας και άκουσα πριν από λίγο ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Ναι, ε, προφανώς όλοι συμφωνούμε στο γεγονός ότι η αρχή της επικουρικότητας ε, ισχύει και προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Δηλαδή, ε, αυτό το οποίο δεν καταφέρνουμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο πρέπει να το κάνουμε σε υπερεθνικό επίπεδο. Δεν, ε, δεν παίζουμε τι λέξει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε απαιτεί να εγκριθούν πολιτικέ, ιδιαίτερα προ την κατεύθυνση τη ανάπτυξη, που ε, δεν μπορούν ε, ε, αυτή τη στιγμή να ασκηθούν σε υπερεθνικό επίπεδο. Ακριβώ γι' αυτό είπε ο πρόεδρο Λαμασούρ το γεγονό ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε ε, την εμπειρία αυτή όπου ε, τα πιο ισχυρά εντό εισαγωγικών εθνικά κράτη, ε, να βάλω και την Ιταλία, αν θέλετε να πούμε τα λιγότερα δύναμα κράτη, έτσι, δεν κατάφεραν να πετύχουν ρυθμούς ανάπτυξης που να έστω να πλησιάζουν κάπως του, του, τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν αλλού. Αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να σκεφτούμε και να αντιλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα. Και εγώ πιστεύω ότι αν κάπου μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα ε, ε, για το ότι τα, τα, ε, τα, τα παλιά κράτη μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους σε διεθνές επίπεδο, κοιτάξτε, αυτό πλέον είναι πόθος, είναι, είναι ψευδέστηση, δεν ισχύει για κανέναν πλέον αυτή η ελπίδα. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε κάτω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε κοινοτικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί είναι προφανές ότι και βεβαίω ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Ε, το στόχο της, ε, της, ε, να φτάσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο ανάπτυξης ανάλογο με τα επίπεδα ανάπτυξης των άλλων. Ε, και βεβαίω, ε, ναι, εξυγίανση των, ε, των προπολογισμών σε εθνικό επίπεδο, βεβαίω, όλα αυτά σωστά, αλλά είδαμε και, τα αποτελέσματα της μελέτης και κοιτάξτε τι να σας πω ενώ ε, μπορούμε να τα μελετάμε, αλλά ξέρετε, έχουμε και μια παροιμία στη γλώσσα μου, τα τελικά, που λέει ότι ε, ενώ σκέφτεται ο γιατρό, ο ασθενή πεθαίνει στο μεταξύ. Τον χάσαμε τον άρρωστο. Αυτή, λοιπόν, ε, αυτό λοιπόν είναι ένα, κάτι, το πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις κρίσης ε, που ε, παρουσιάζονται και η τελευταία κρίση της Ελλάδας, η πρόσφατη κρίση της Ελλάδας θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί ως δίδαγμα. Ε, τα συμπεράσματα της ε, μελέτης ε, που μας παρουσιάσατε σήμερα ε, ακόμα και ρίχνοντας, ε, μα οδηγούν στο εξή, ότι ακόμα και μία ματιά να ρίξουμε στον προπολογισμό ε, για το 2011, ε, μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πραγματικά θα πρέπει ε, να, λάβουμε, να, να δούμε ε, τι γίνεται ε, αλλά, ε, και, τι, και, είναι, και ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνοντα υπόψη τους δημοσιονομικούς προ, προϋπολογισμούς και τους ιδίους πόρους. Ε, και, και ακριβώς όλα αυτά εξηγούν το πόσο μικρή είναι η συμβολή της σε, σε κοινωτικό επίπεδο. και όπως είπε και ο συνάδελφος, τα, περισσότερα, τα περισσότερα χρήματα και οι περισσότερες αποφάσεις δεν, δεν αφορούν αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τους, αλλά τα επιμέρου κράτη. Αυτά όμω ε, έχουν να κάνουν και με το εξή. Ε, και με την κοινή γνώμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ε, αντιλήφθηκε την ανεπάρκεια δυνατότητας μιας ισχυρής απάντησης της Ευρώπης για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αλλά και το ζήτημα της ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, είναι αναπόφευκτο ε, να ξαναρχόμαστε στο παλιό ερώτημα το οποίο το έθεσε και ο κύριος Λαμασούρ αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή να δούμε κατά πόσον διαθέτει επαρκή πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση των στόχων της. Και ορισμένοι στόχοι δεν, δεν μπορούν να, να υλοποιηθούν αλλιώς παρά μόνο σε εθνικό επίπεδο. Το είπα και πριν από λίγο. Άρα λοιπόν, για, στην πορεία προ την ολοκλήρωση θα πρέπει να έχει και οικονομικά και δημοσιονομικά μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή τη για να απαντήσει στι προκλήσει των καιρών αλλά και στι προσδοκίε των πολιτών. Γιατί, ε, όπω είπαμε και πριν από λίγο, οι, ε, είδαν οι πολίτε ε, την ανάγκη ύπαρξης ενός πραγματικού ε, ε, ελέγχου, δημοκρατικού ελέγχου που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος συντονισμό ανάμεσα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και στου εθνικούς προπολογισμού, τουλάχιστον εν μέρη, θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτές τις προσδοκίες, σε αυτέ τις απαιτήσει. Και γι' αυτό ακριβώ σα είπα ότι βρίσκω θετική αυτή την ιδέα που ακούσαμε. Και θα πρέπει βεβαίως ε, ε να, δούμε ε, πώς ακριβώς θα κάνουμε αυτή τη σύγκριση των εθνικών προϋπολογισμών με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια κατάρτισης των υπολογισμών θα πρέπει να είναι ομοιογενή ε, για να μπορούμε ε, να συγκρίνουμε με, με αντικειμενικό τρόπο τα στοιχεία. Εμεί, κοιτάξτε, προσπαθούμε να το κάνουμε και σε εθνικό επίπεδο αυτό. Να δούμε δηλαδή τον εθνικό προπολογισμό σε σχέση με του περιφερειακού προπολογισμού. Ε, ε, για να μπορέσουμε λοιπόν, να κάνουμε μία σύγκριση, ε, χρειαζόμαστε ε, ομοιογένεια ανάμεσα στους εθνικο, στον εθνικό ε, προπολογισμό και στου περιφερειακού. Ε, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και τη λογική του φεντεραλισμού και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε αναλογία και σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω κύριε Λαμασούρο ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία ακούσαμε εδώ. Ε, τόσο όσον αφορά μια κοινή συζήτηση, εγώ έτσι θα την ονομάσω, για τους προπολογισμού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα, ε, ε, ε θα, θα, δούμε το ζήτημα ε, του κεντρικού ρόλου του Κοινοβουλίου, του δημοκρατικού ρόλου λοιπόν που μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναντι πολιτικών που στη συνέχεια θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο και συμφωνώ ταυτόχρονα και με αυτή την διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη για ε, τη διεξαγωγή αυτών των συζητήσεων και των προβληματισμών. Υπό το βλέμμα των άλλων λοιπόν, έτσι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια γιατί ε, και, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν αρμοδιότητε επί του προπολογισμού. Αυτή η συνδιάσκεψη λοιπόν πιστεύω ότι θα επιτρέψει για τον καλύτερο προσανατολισμό ε, των ε, συζητήσεων για τι βασικέ επιλογέ ε, προπολογισμού και, και σε επίπεδο Ευρώπη αλλά και σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων. Και τέλος, συμφωνώ και με αυτή την Ευρωπαϊκή Οικονομική ε, Διάσκεψη ε, που, ε, με πρωτοβουλία της επόμενης Προεδρίας της Βελγικής για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον καταμερισμό των ρόλων των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, για το σύστημα των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον συνολικό έλεγχο. Και κλείνω λέγοντάς σας ότι εγώ πιστεύω ότι ε, όποιο έχει αυτή την αυταπάτη, ότι δηλαδή περισσότερο συντονισμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια θα μας οδηγήσει, ε, θα οδηγήσει σε. Ε, ε, θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, να σα πω το εξή. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά ε, τι ε, πιστώσει του ευρωπαϊκού προπολογισμού, αυτό αποτελεί μοχλό και για τις εθνικές επενδύσεις ε, και κυρίως για τις ιδιωτικές επενδύσεις ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεύτερον, οι δημόσιε δαπάνε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητε για την επίτευξη, με βάση την αρχή τη επικουρικότητα, την οποία αναφέρθηκε και πριν από λίγο, επίτευξη λοιπόν στόχων, ε, υψηλών στόχων, υψηλή προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που δεν μπορούν να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο. Οι νέε προτεραιότητε, στρατηγικέ προτεραιότητε που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία κτλ. Ή το θέμα τη μετανάστευση, το ίδιο το θέμα τη μετανάστευση. Και εμεί στην Ιταλία ε, μα πονάει το θέμα αυτό. Ε, γιατί είμαστε μια, θάλασσα που ε, είμαστε μια χώρα που πρέχεται από παντού από τη θάλασσα και καταλαβαίνετε ότι δεχόμαστε από παντού μετανάστες. Τρίτον, ε, και αυτό ε, είναι η δική μου ε, ε, άποψη με όλη τη μετριοπάθεια για το θέμα της ολοκλήρωσης, της περισσότερης ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ χρειαζόμαστε μια παρέμβαση σε επίπεδο προπολογισμού της Ευρώπης, ισχυρή παρέμβαση που να είναι ορατή από τους πολίτες. Άρα λοιπόν ε, δέσμευση πόρων και κονδυλίων σε έργα με υψηλή ευρωπαϊκή ε, προστιθέμενη αξία. Αριστεία των πανεπιστημίων, υγεία, υποδομές. Ε, να δείξουμε δηλαδή συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής δράσης. Να δείξουμε ότι με την Ευρώπη τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα από αυτή την κρίση να μπορέσουμε να δράξουμε την ευκαιρία και να την μετατρέψουμε σε μια θετική εμπειρία. Και αυτό δεν σα τα λέω με, με κάποια ρομαντική διάθεση. Ελπίζω να σα πείσω όλου ε, για αυτό το οποίο είπε και ο πρόεδρο Λαμασούρ. Για το ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει τη δίαιτα ε, τη δίαιτα δυνατίσματος που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, τη λιτότητα. Ε, ο συντονισμός λοιπόν ανάμεσα στους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς και, ε, και, στο, και, στο, Ευρωπαϊκό Κοινοβου, και στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι προς συμφέρον όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε χυμαρόδος παράβαση. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα. Και ιδιαίτερως αναφερθήκατε σε μια από τις συστάσεις της Deloitte για ένα σύστημα ενοποίησης των ε, δημοσιονομικών, εθνικών και ευρωπαϊκών και περιφερειακών κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να κριθεί το αλγευρικό άθροισμα των εθνικών μας προϋπολογισμών και ο αντίκτυπός τους στις οικονομικές μας πολιτικές. Αν θέλουμε να κρίνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των οικονομικών μας πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με αυτά της Βραζιλίας, της, ε, των Πολιτειών κλπ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ε, συμπίληση τέτοιων είδων από τέτοιου είδου αποτελεσμάτων. Ο κύριος Γκέρεν μεταξύ έχει στήσει το λόγο εδώ και λίγη ώρα και έστω συγγνώμη που τον καθυστέρησα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποδεικνύεται, έστω και με κάποια καθυστέρηση, ότι η υγεία του ατόμου ορίζει τη δημόσια υγεία, την υγεία του όλου. Αυτό βλέπουμε στα δημοσιονομικά της Ευρώπης και πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Μετά από την ε, πρόταση του Ρεν και του Μπαρόσο, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται και η ειλικρίνεια φυσικά και γι' αυτό θα ήθελα και έχω να πόσο κάποιες προτάσεις σχέσεις με τις δικές σας ιδέες για την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στο διάλογο που προηγείται της έγκρισης των προϋπολογισμών. Για να μην χάνουμε χρόνο λοιπόν, φρονώ ότι καλό θα ήταν προκαταβολικά, καταρχά βέβαια πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξη τη πρόταση, αλλά και επίσης προκαταβολικά να ε, καταγράψουμε το τι θα μπορούσε να είναι ενοχλητικό σε, αυτή την, ε, σε αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή, να δούμε πού υπάρχουν ε, παραθυράκια, μέθοδοι απόκρυψης, κρίζες ζώνες, εκεί δηλαδή που ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να αποκρύπτουν την δημοσιονομική του υγεία, τα κράτη-μέλη από τους εταίρους τους, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό νομίζω ότι όσοι έχουν δεχθεί, εγκρίνει το σύμφωνο σταθερότητας, είναι υποχρεωμένοι να, να τηρούν καθαρά και διάφανα δημοσιονομικά. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς τώρα με το screening ε, να ισχυριστεί ότι υποχρεούται να εγκαταλείψει ηθική του ε, κυριαρχία ή τις ε, επιλογές τις εθνικές. Όχι, δεν πρόκειται περί εθνικής κυριαρχίας, πρόκειται μόνο από, συν... από παράγοντα που απορρέει από το σύμφωνο σταθερότητα. Είναι πολύ απλό. Θέλετε αυτή την αρχή, ναι. Ε, απόρρια της αρχής είναι ο έλεγχος και έλεγχος εκ των προτέρων που μπορεί να αποβεί και χρήσιμος ώστε να αποφευχθούν και οι περιπτώσεις απόκρυψης και να προσδιοριστούν βέβαια ε, τα όρια δράσης των κρατών Και νομίζω θα μπορούσαμε να προβάλλουμε και ένα δεύτερο επιχείρημα, ώστε να πούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν χάνουν προνόμια οι αρμοδιότητες των αντίων βγαίνουν κερδισμένα γιατί από τη διαδικασία προτείνατε εσείς αν την εννοώσα σωστά, και οι 27 και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν εκ των προτέρων δικαίωμα εξέτασης των δημοσιονομικών διαδικασιών που προκύπτουν ε, σε άλλα κράτη-μέλη. Και καθώς όλοι υποχρεούμεθα να ακολουθούμε την δημοσιονομική πειθαρχία, είναι αυτονόητη αυτή η υποχρέωση, μάλλον το δικαίωμα εξέτασης προκαταβολικής των δημοσιονομικών των άλλων. Επίσης, Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό το screening, αυτή η εξέταση θα πρέπει να, έχει να, να επεκτείνεται όχι μόνο στη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και στην ανταγωνιστικότητα. Και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα να συζητήσουμε μεταξύ μας έτσι ώστε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να είναι ωφέλιμη, να αποβαίνει εις όφελο των πάντων. Και επίσης τελευταία παρατήρηση καλό θα ήταν να σταματήσουν οι παράτερες και Αντιφατικέ απόψει που αποφέρουν ει βάρο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά του ευρώ. Για να κάνει κανεί φάλσο συνήθω χρειάζεται να παίζουν διάφορα όργανα. Βλέπουμε όμω ότι ορισμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν καταφέρει με πολύ ε, ανεπτυγμένο ταλέντο πρέπει να πω μόνοι του να αποτελούν φαλ, ε, ορχήστρα που φαλτσάρει ταυτόχρονα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ορισμένοι των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έχουν ακολουθήσει δηλώσεις, τη μία στο άσπρο και την άλλη στο μαύρο, που είναι απολύτως αντιφετικές μεταξύ τους. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Πρέπει να πω ότι εκτιμώ την ειλικρίνειά σας. Ε, you speak plainly, όπως λένε οι Άγγλοι. Και δεν χρησιμοποιείτε ξύλινη γλώσσα. Ε, θίγεται ένα θέμα και έχετε το θάρρος να το θίξετε. Ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν συζητούμε πολύ μεταξύ μας όταν λέτε ότι πρέπει να, ε, να, ερευνήσουμε τις υπεκφυγές και αυτό έγινε προετών στη χώρα μου. Εγώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι την εποχή που ήμουν υπουργό η Γαλλία ήταν άμεμπτη ως προς τις πληροφορίες που έστελνε στις Βρυξέλλες. Ελπίζω ότι τώρα όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή, αυτό το οποίο ενδεχομένως φάνηκε κραυγαλαία στην περίπτωση της Ελλάδος μπορεί να ισχύει και να υπάρχει και, παλού, και αλλού διότι εν τη σοφία τους τη δεκαετία του 1980 οι τότε πολιτικοί θύνοντες αποφάσισαν να συμπληρώσουν τους κοινοτικούς πόρους από εθνικές συνδρομές οι οποίες θα ήταν αντίστοιχες του πλούτου κάθε χώρας δεν είναι τυχαίο ότι πήρανε το ΑΕΠ σαν βασικό κριτήριο πήραν σαν βασικό κριτήριο για να ε, αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν τον πλούτο κάθε χώρας τη βάση ε, ε, του ΦΠΑ και το ΑΕΠ θεωρήθηκε συμπλήρωμα και έκτοτε από την ε, εποχή εκείνη έχει γίνει πρόοδος ως προς την αξιολόγηση των διαφόρων χωρών γίνονται και οι μελέτες του Eurostat αλλά υπάρχουν ακόμη δυνατότητες ερμηνείες και σε ορισμένες χώρες υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες συγκεντρώσεως πληροφοριών μπορεί σε ορισμένα σημεία να υπάρχει ο πειρασμός να μην τα πει όλα στις Βρυξέλλες και αυτά είναι που θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να θίξουμε σαν θέματα. Και γι' αυτό ο πρόεδρος Βαν Ρομπόη σκοπεύει ε, στα πλαίσια ε, της, ε, σκοπεύει να πράξει στα πλαίσια της αποστολής που του έχει ανατεθεί. Θα θέλω τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μοταπίλ από την Πορτογαλία. Σα ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε γιατί διοργανώσατε αυτή τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ήθελα να σας πω ότι στο Κοινοβούλιο μου το θέμα αυτό ε, συζητείται από την Επιτροπή Προπολογισμών και από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ε, όσον αφορά λοιπόν αυτή τη συζήτηση και το συντονισμό ε, με, τον, ε, με το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό σας λέω ότι αυτό θα συζητηθεί ε, είναι θέμα το οποίο ε, συζητείται και από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έτσι, στη χώρα μου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα αυτό πρέπει να σας πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούσαμε και είπατε συμφωνώ και με τις υποδείξεις αυτές νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει είναι εμφανές ότι θα πρέπει να συντονίσουμε τις πολιτικές μας τις δημοσιονομικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο με την ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Πράγματι, ε, χρειαζόμαστε μία ανάλυση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη ε, συμβολή ε, της Ευρώπης για την επίτευξη των πολιτικών και των στόχων. Καθώς επίσης να δούμε και σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να αναπτύσσονται αυτές οι πολιτικές αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των χωρών μας. Κοιτάξτε, δεν έχω λάβει εντολή να σας πω κάτι σε σχέση με τον εκ των προτέρων έλεγχο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι και το θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ε, σήμερα. Ε, πιστεύω όμως ότι η πρόταση για μια κοινή συζήτηση, για μια ημερίδα είναι πάρα πολύ καλή. Ε, τώρα, πρέπει να καταλάβουμε υπόψη ότι ε, οι, μακροοικονομικέ μακροοικονομικές ε, δημοσιονομικές προοπτικές είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Εμένα μου δημιουργεί έκπληξη το γεγονός ότι ε, το γεγονός ότι ακολουθούμε μια άλλη οδό σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε τα πλαίσια για τη σύγκριση των εθνικών προπολογισμών. Και εδώ συμπεριλαμβάνω αυτό το οποίο θα ονόμαζα περίμετρο του προϋπολογισμού, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε ε, να συγκρίνουμε ε, τα διάφορα επιμέρους στοιχεία και το πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα στοιχεία τα οποία είναι και καλυμμένα κατά κάποιο τρόπο. Ε, πολύ καλή λοιπόν αυτή η ιδέα για εκείνη τη συζήτηση και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν και τα εθνικά κοινοβούλια να καταλάβουν καλύτερα και τις τεχνικές πτυχές του ζητήματος. Πάντως στην Επιτροπή που είμαι πρόεδρος αντιλαμβανόμαστε ότι μερικές φορές συζητήσεις δεν είναι πολιτικής φύσεως αλλά τεχνικής φύσεως ε, συγκρισιμότητα, αλλαγή μεθοδολογίας ε, ε, μέθοδο υπολογισμού κτλ. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτή ε, η προσπάθεια που γίνεται στην ε, Πορτογαλία ε, σε, και σε τεχνικό επίπεδο για να δούμε πώς μπορεί να μειωθεί το δημόσιο χρέο. Ε, αυτή η προσπάθεια λοιπόν δική μας σε επίπεδο θα μπορούσε να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί και από την κοινή αυτή συζήτηση. Και θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τις εκθέσεις δημοσιονομικού προσανατολισμού. Όλα αυτά πάντως βεβαίως θα πρέπει να στηρίζονται σε μια ανταλλαγή στοιχείων και απόψεων. Βεβαίω, ε, δεν αναφέρομαι μόνο στις εκθέσεις ε, προσανατολισμού των προπολογισμών. Και κάτι άλλο. Ε, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα ε, είναι ε, να δούμε ε, τη σχέση των εθνικών δράσεων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, και, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει, και αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να βοηθήσει τα εθνικά κοινοβούλια κατά την αξιολόγηση των δικών τους προπολογισμών. Και βεβαίως υπάρχει μερικές φορές αυτή η διαφορά ανάμεσα στον μονοετή προπολογισμό και στον πολιετή που ακολουθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κοιτάξτε, τα προγράμματα, τα, τα προγράμματα ανάπτυξης σταθερότητας που πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη έχουν ήδη πολιετή προγραμματισμό. Άρα και αυτό δεν είναι πρόβλημα επί της ουσίας. Με δύο λόγια συμφωνώ με αυτή τη μεθοδολογία την διακοινοβουλευτική ε, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαφάνεια ε, και ως προς τον συντονισμό των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και επειδή θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούν τα, τα Εθνικά Κοινοβούλια για τη σύγκριση των ε, προπολογισμό τους με τον προπολογισμό των άλλων. Επίση, να ξεκαθαρίσουν καλύτερα τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ε, δίνει το λόγο στην Έλγια Τρίπελ από την ομάδα των Πρασίνων για να υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ Βορράς και Νότου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω με την, κατάθεση της, στη, με την κατάσταση της κρίσης που βρισκόμαστε. Έχουμε ένα θέμα σταθερότερο του ευρώ όπου θέτει μία νέα πρόκληση. Έχουμε την οικονομική κρίση και την κρίση των χρηματαγορών που οφείλονται σε λάθη. Γι' αυτό και υπάρχει η κρίση Πρέπει λοιπόν να υπάρξει το πολιτικό θάρρος να διδαχθούμε από τα λάθη μας και να αναρωτηθούμε τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε διότι ε, το γραφείο μας είπε ότι υπήρξαν λάθη στη στρατηγική της Λισαβόνας. Δεν υπήρχαν εστιασμένες δράσεις στον προϋπολογισμό ο κατά τρόπον ώστε οι στόχοι τους οποίους είχαμε διατυπώσει πραγματικά να εφαρμοστούν. Τι διδασκόμαστε από αυτό, ποια είναι η δημοσιονομική πολιτική η οποία πρέπει να συνδυαστεί με τους πολιτικούς μας στόχους και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη διότι διαφορετικά αυτό το οποίο έγινε ε, πριν 10 ε, χρόνια τις, με τη στρατηγική της Λισαβόνας για το 2020 δεν θα υλοποιηθεί και θα ξαναναρωτιόμαστε πάλι πού βρισκόμαστε στο μέλλον. Οπότε ε, κύριε Λαμασούρ εσείς αναφέρατε την ασθενή ανάπτυξη στη Γαλλία, στη Γερμανία που είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στην Κίνα, στην Αφρική και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας λυπεί αυτή τη στιγμή αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε ε, τα πρότυπα αναπτύξεως πριν από το 2007 αυτά τα οποία εφαρμοζόντουσαν ήταν σωστά πρότυπα αναπτύξεως. Ε, αν ξεκινήσουμε από αυτό το σκεπτικό και από την οικονομία χαμηλού διοξιδίου του άνθρακος βλέπουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις θεωρήσεις μας και να δημιουργήσουμε μία νέα μέθοδο όσον αφορά την τεχνολογία, τα βιώσιμα καύσιμα για να μπορούμε να έχουμε μία κοινωνία με μικρότερη ανάπτυξη και νομίζω ότι αυτό θέλω να ρωτήσω και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εάν ξεκινήσουμε από τον τίτλο της συνεδριάσεως να δημιουργηθούν μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών πρέπει να αναρωτηθούμε αν έχουμε την πολιτική δύναμη για να εντοπίσουμε τους οικονομικούς στόχους για να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη της για τα επόμενα έτη. Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν δεν το επιτύχουμε, αν δεν εντοπίσουμε τα κοινά πολιτικά συμφέροντά μας, τότε ο καυγάς ο οποίος έχει ξεκινήσει θα διαιωνίζεται. Και γι' αυτό ξεκινώ από αυτά τα οποία ελέγχθησαν σήμερα το πρωί και θα ήθελα να θίξω ορισμένα θέματα τα οποία μπορούν να προσφερθούν για εφαρμογή κοινή πολιτικής. Παραδείγματο χάρη οι δαπάνες για την ε, ε, εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την έρευνα για όλα αυτά που τώρα λέγονται ε, μία πολιτική προσαρμογή σε μία οικονομία που δεν θα χρησιμοποιεί ε, τον άνθρακα και το διοξίδιο του άνθρακος όπου θα πρέπει να υπάρξουν συνολικές λύσεις διότι τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από την Κίνα και από τις Ηνωμένε Πολιτείες και να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προτέρημα. Άρα από πού προέρχονται ε, οι δυνάμεις μας. Προφανώς όχι από το να διαιωνίσουμε αυτό που κάναμε τα δέκα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης και πρέπει να κάνουμε κάτι νέο και συγχρόνως θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους οικολογικούς μας στόχους και ελπίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε και του άλλες υπήρους να μας ακολουθήσουν ακολουθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης όσον αφορά την εσωτερική αγορά αλλά και την παγκόσμια οικονομία, τα θέματα της νεολαίας, της εκπαιδεύσεως, της έρευνας, της βιώσιμης ανάπτυξης, πώς τα θέματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν κατά τρόπον ώστε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί για την Ευρώπη του 2020 στο χαρτί να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερες τέτοιες ε, κοινέ συνεδριάσεις για να δούμε αν υπάρχουν πολλά κοινά συμφέροντα που μπορούν να διαγραφούν και να εντοπιστούν μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά τρόπον ώστε οι στόχοι μας αυτοί να μπορέσουν να επανδρωθούν με πόρους και να υλοποιηθούν. Το θέμα ακόμη αμφισβητείται, αλλά χωρίς να υπάρχει μία κοινή προσπάθεια και κοινά συμφέροντα τα οποία θα ε, εντοπιστούν δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μία ποιοτική βελτίωση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Παπανδρέου, παρακαλώ, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να σας συγχαρώ για τη σημερινή συζήτηση και τις προτάσεις και νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτές οι συναντήσεις να γίνουν πιο συχνές μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για και ενημέρωση αλλά και συντονισμό των ενεργειών μας γιατί πολλές φορές υπάρχει ανταγωνιστικότητα ή αντίθεση ε, λόγω έλλειψης ε, γνώσης. Ε, το τι κάνει ο κάθε φορέας Εθνικό Κοινοβούλιο ή Ευρωκοινοβούλιο, το τι πολιτικές ακολουθεί και το τι προτεραιότητες ε, βάζει. Ε, η έκθεση της Επιτροπής σας νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την, ε, στην προσπάθεια να αναλυθούν τα αίτια της μειωμένης <clears throat> συνέργειας μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Εθνικών Προϋπολογισμών και του Κοινοτικού. Ε, είναι γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς όπως η έρευνα και η τεχνολογία που αναφέρεται η συνέργεια είναι μεγαλύτερη και αυτό ίσως επειδή υπάρχουν και οι χρηματικοί πόροι οι οποίοι με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα που υπάρχει καλύτερο συντονισμός και καλύτερο αποτέλεσμα όπως επίσης και σε θέματα εξωτερικής βοήθειας λόγω της εκχώρησης ε, εκ μέρου των εθνικών ε, ε, των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την και με αυτόν τον τρόπο έχουμε οικονομίες κλίμακος. Ενώ σε άλλους τομείς η συνέργεια δεν είναι τόσο αποτελεσματική, διότι είτε τα, η συμμετοχή του ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε ορισμένες χώρες είναι πολύ μικρή και άρα δεν υπάρχει κίνητρο για να συντονίσουν τις ενέργειες, είτε γιατί οι πολιτικές ε, ασκούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι είναι τώρα μια ευκαιρία μετά την οικονομική κρίση και τα προβλήματα τα οποία έχουμε ε, μάλλον σας ακούω λίγο αισιόδοξο για το ε, ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης. Ελπίζω να δικαιωθείτε. Ε, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη ότι έχουμε ξεπεράσει ως Ευρώπη, ως παγκόσμια οικονομία τα πολύ δύσκολα και γι' αυτό χρειάζεται καλύτερο συντονισμός και συνεργασία μεταξύ μας. Επίσης έχουμε την μία επιτυχία, για να μην πω αποτυχία, τη στρατηγική της Λισαβόνας και ίσως είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλα τα διδάγματα το τι έφτεξε και το τι πρέπει να γίνει για να ξεπεράσουμε και τις δυσκολίες αλλά και για να δημιουργήσουμε τους θεσμούς τις πολιτικές, τους κανόνες και τις κυρώσεις που είναι απαραίτητες ώστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι η συζήτηση και η συνέργεια μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητο για μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, διαφάνεια είναι ζητούμενο πλέον σε, όλες, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πολιτικές και τους θεσμούς, τη λειτουργία των θεσμών και θα πρότεινα εκτός από την πρότασή σας η οποία είναι πάρα πολύ σωστή και, και συμφωνώ ε, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει ευθυγράμμιση των κατηγοριών των δαπανών προϋπολογισμού σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και η Eurostat θα μπορούσε να διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ εθνικών και κοινοτικών δημοσίων δαπανών και να προβεί σε συγκεντρωτική ανάλυση των ευρωπαϊκών δημόσιων οικονομικών. Θα πρέπει επίσης οι στόχοι και οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλαμβάνονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών και αυτό θα επιτρέψει τη σύνδεση των εθνικών στόχων με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αποτέλεσμα την ε, δημιουργία ενός πλαισίου που θα επέτρεπε τη συνύπαρξη κοινοτικών και εθνικών ε, δαπανών και βεβαίω χρειάζεται ένα απαραίτητο μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε όμω, κύριε Πρόεδρε, να μην ξεχνάμε το γεγονό ότι σήμερα ε, όλο και περισσότερε χώρε αναγκάζονται, παρόλο που έχουν ε, το, τα προγράμματα ε, ε για την δημοσιονομική πειθαρχία προγράμματα ανάπτυξης και σταθερότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά, αναγκάζονται ορισμένε φορές να παίρνουν έκτακτα μέτρα για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή κάποιων αποκλήσεων. Ε, και αυτό επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα περιθώρια ελιγμών στην άσκηση πολιτικής και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ εθνικών και κοινοτικού προϋπολογισμού. Πάντως νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη και συζήτηση και ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συμφωνήσω μαζί σας οι συναντήσεις αυτές να γίνουν πιο συχνές ε, και όχι μία φορά το χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Παπανδρέου. Σημειώνω ιδιαίτερος ότι και εσείς εκφράσατε την επιθυμία για πιο αξιόπιστα μέσα ισολογιστικά, αλλά και συγκρίσεις πιο ευχαίρεις μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πρόκειται για μια από τις συστάσεις του γραφείου Deloitte. Ε, μια παρατήρηση. Όλοι με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε τόσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Θαυμάζουμε την παρεσία των ελληνικών αρχών, οι οποίες ε, ε, καταρτίζουν και εφαρμόζουν μια πολύ αυστηρή πολιτική δημοσιονομική που είναι δύσκολο να δεχθεί και ο λαός προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα να ανακάμψει από την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής οικογένειας και όχι των επιμέρους αλληλεγγύων μεταξύ εθνών ή κρατών. Εάν περιοριστούμε στην διακρατική στήριξη, όταν τα πράγματα πάνε πράγματι πολύ άσχημα, έχουμε την αντιπαράθεση τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών. Και εν προκειμένου στην κρίση αυτή ακούστηκαν εκάστοτε σοβινιστικού ακόμη τύπου ε, προκαταλήψεις εις βάρος κάποιων κρατών, προκαταλήψεις χαρακτήρα που δεν έχουμε δει εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπη. Ενώ τον αντίον, εάν προβάλλουμε την αλληλεγγύη, την ευρωπαϊκή, την αλληλεγγύη της οικογένειας, οπότε ο ένας εξημών πάει, τα, τα έχει κάπως πιο δύσκολα και η ζωή αυτά φέρνει. Σήμερα είναι η Ελλάδα, μεθαύριο θα είναι κάποια άλλη χώρα από τις δικές μας. Εάν λοιπόν όλη, βοηθη, όλη, όλη η οικογένεια σταθεί στο πλευρό του, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ενώ εάν πούμε, για να δούμε, ένας από την οικογένεια έχει δυσκολίες, ποιος από εμά θα πάει να τον βοηθήσει και για πόσα, πόσα θα του δώσουμε δηλαδή να πάει να βοηθήσει, τότε είναι πολύ πιο δυσχερή η λήψη της απόφασης και προφανώς προκαλούνται και ε, εντάσεις όλο το, ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ακριβώς το στόχο αυτό έχει να ε, εξουδετερώσει τις εντάσεις. Φυσικά δεν μπορούμε κάθε ένταση, κάθε ε, διαφοροποίηση, κάθε αντίθεση μέσα στο διάλογο να την ε, εξουδετερώσουμε γιατί αυτό Άλλωστε προποθέτει και η δημοκρατία. Αλλά πάντω μπορεί να καλύψει, μπορεί να δώσει διέξοδο το εντάσει έτσι ώστε να βοηθηθεί και μια χώρα να βγει από την κρίση. Α ξαναπεράσουμε λοιπόν στη βόρεια Ευρώπη με την Ιζαμπέλ Τζιρόν που εκπροσωπεί την προσεχή Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά είπατε, ξεκινώντας, ότι μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι είμαστε παράλληλοι κόσμοι, δεν έχουμε δηλαδή φυσικές, φυσιολογικές σχέσεις και θα πρέπει να, καταβληθούν, ε, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συναντηθούμε και να συναντιόμαστε τα εθνικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, φάση της προετοιμασίας και της χάραξης των μεγάλων παραμέτρων ε, για όλα τα κύρια οικονομικά ζητήματα. Και για να επανέλθω στα όσα είπε ο συνάδελφο Ρεν, θα ήθελα να μιλήσω και για τα εθνικά κοινοβούλια και τα μέσα που θα πρέπει να του προσδώσουμε για να αντιμετωπίσουμε, δεν θα πω εγώ τη λέξη παραθυράκια, αλλά την παραχάραξη των ε, υπουργών τη ε, της εθνικής οικονομίας γιατί και εγώ έχω διατελέσει υπουργό οικονομικών και ξέρω πολύ καλά πως μέσα από και υπό την κάλυψη της ευρωπαϊκής ομπρέλας αλλά και με κάποιο είδους παραχάραξη των δημοσιονομικών μπορούμε να παρουσιάσουμε στοιχεία τα οποία είναι αδιαφανή και μη πρόσφορα στον έλεγχο. Σε αυτά λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ελέγχου στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια εναντί των ε, Υπουργών της Εθνικής Οικονομίας που υποβάλλουν τον προπολισμό αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενάντια της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Πέραν αυτού αλλά και με τον στόχο μιας ευρωπαϊκής ανάπτυξης αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, πιο ποιοτικής ανάπτυξης όπως αυτή που περιέγραψε στην Άλφος πέρι πολύ σωστά, πρέπει να επιβάλλουμε πειθαρχία στα κράτη-μέλη και ο δημοσιονομικός συντονισμός είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος πιστεύω, διότι πέραν αυτού του δημοσιονομικού συντονισμού τίθεται το ζήτημα του ε, φορολογικού συντονισμού και ξέρω ότι το ζήτημα είναι ακανθώδες, ναι βεβαίως, θα πρέπει να το συζητήσουμε όμως. Δεν έχει νόημα δηλαδή να επικεντρωθούμε μόνο στο δημοσιονομικό συντονισμό, εάν δεν κοιτάξουμε και τη φορολογική όψη, γιατί η έκθεση Μόντι μίλησε για την ε, προοπτική την ευρωπαϊκή, αν δεν υπάρξει καλύτερο συντονισμό ω προ το ΦΠΑ, το φορολογικό, τη φορολογική μεταχείριση του περιβάλλοντο, δηλαδή τον περιβαλλοντικό χώρο, την φορολογία ή τις βασικές αρχές φορολόγησης των ε, ιδιωτών ε, ή των νομικών προσώπων. Και υπάρχει βέβαια ζήτημα και συντονισμού όχι μόνο της φορολογίας αλλά και του χρέους, δηλαδή επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο μέρος ή τμήμα της αγοράς ε, έχει πρόσβαση στον εθνικό πλούτο. Και αυτό μέσα από μια πολιτική ε, που θα σήμαινε για τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα και συμμετοχή στη χρηματοδότηση των μεγάλων ε, διευρωπαϊκών σχεδίων, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το Γαλιλαίο κτλ. Και όπω είπε και ο Πολωνός συνάδελφο, μια άλλη η εικόνα θα ήταν να ε, στηρίζει το ένα κράτος το άλλο όταν έχουμε στήματα μάλλον να υπάρχει συντονισμένη στήριξη των κρατών ε, που πλήττονται από φυσικές καταστροφέ πλημμύρες κτλ. Τα αισθήματα της εκπαίδευση, της επιμόρφωσης θα πρέπει να δούμε αν τηρούνται οι στόχοι που ορίζονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και από τους εθνικού προπολογισμού. Και επίσης η λεγόμενη βελγική συνθήκη, δηλαδή η συνθήκη σχετική με την ρύθμιση των δημοσιονομικών στο Βέλγιο, και πρέπει να σας πω ότι ναι, εγώ ανήκω μεν στην αντιπολίτευση στην πατρίδα μου, αλλά θα υποστηρίξω κάθε λύση η οποία θα πρότεινε μία προοπτική συνθήκης η διαπραγμάτευσης για τα θέματα τα δημοσιονομικά με προσθήκη και των βασικών θεμάτων εκείνων που χρειάζεται από κοινού να επιληθούν, ώστε να έχουμε όχι μόνο στη δημοσιονομική και οικονομική πτυχή, αλλά και γενικότερα με περισσότερη συνοχή και συντονισμό που είναι όλο και πιο απαραίτητος. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Ιζαμπέλ και ως ήθιστε Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από Βελγική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι, όπως ξέρεις, έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Βέλγιο. Δεν ξέρω αν οι Βέλγοι έχουν εμπιστοσύνη στο Βέλγιο, αλλά εμείς περιμένουμε πολλά. Και κάθε φορά που ε, εναλλάσσεις την Προεδρία του Βέλγιο, ξέρουμε ότι παίρνει βήματα, παίρνει μέτρα που επιταχύνουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ας γυρίσουμε τώρα προς τα νότια και τη Ρώμη με τον Τζαν Καρλο Τζότζα, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ. Το σημερινό θέμα το οποίο μας απασχολεί αφορά το συντονισμό ανάμεσα ε, στις ε, Εθνικές Επιτροπές Προϋπολογισμού ε, με, την, με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό θα οδηγήσει σε ε, μια ε, βελτιωμένη συνεργασία στον τομέα αυτό, ε, κυρίως εδώ όπου αυτή τη χρονική στιγμή όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των περικοπών από τη μία και από τη λιτότητα και από την άλλη της ανάπτυξης. Βεβαίως και απαιτείται συντονισμός, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε κοινή γλώσσα. Ε, κοινή γλώσσα ε, σημαίνει ότι όσοι ασχολούνται με θέματα του προπολογισμού ε, θα χρησιμοποιούν ε, εναρμονισμένα στοιχεία, αν θέλετε, για να μπορέσουμε, ε, να, για να, μπορέ, να, είναι, να μπορέσουμε να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία και να αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ε, κοινοτικό. Και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνονται συναντήσεις όπως η σημερινή όπου ε, ε, γίνεται σύγκριση αυτών των αριθμητικών στοιχείων, αλλά και πέραν αυτών γίνεται ένας διάλογος. Το πρόβλημα είναι, κύριε Λαμασούρ, ότι ε, πρέπει να δούμε ε, ε, πώς ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα των εθνικών προϋπολογισμών ταιριάζουν με το χρονοδιάγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερον, όσον αφορά τις ε, διαδικασίες και το είπε και ο συνάδελφος ε, προηγουμένως από την Ιταλία ε, εμείς μεταρρυθμίσαμε την ε, διαδικασία προπολογισμού κυρίως όσον αφορά τον χρονικό προγραμματισμό να δούμε λοιπόν ε, πώς όλα αυτά συνδυάζονται με τις έκτακτες περιστάσεις και με την κρίση ε, συνήθως η διαδικασία του, η συζήτηση του προπολογισμού γίνεται το φθινόπωρο, αλλά η πιο σημαντική συζήτηση ε, γίνεται στις προσεχείς ημέρες, στις προσεχείς εβδομάδες. Ε, όπως άλλωστε γίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το θέμα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το θέμα του χρονικού προγραμματισμού και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να, για να έχουμε έγκαιρες απαντήσεις. Αν θέλουμε σε τελευταία ανάλυση να παίξουμε προσταγωνιστικό ρόλο. Αν δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια είναι έτοιμα να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εξίσου έτοιμο. Γιατί, κοιτάξτε, κατά την απόψή μου, για προφανείς λόγους και για λόγους ε, αποφασιστικής λήψης αποφάσεων, τι αποφάσει παίρνουν κυρίω οι κυβερνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα υπάρχει ο κίνδυνο να αποξενωθούν από την όλη διαδικασία τα εθνικά κοινοβούλια. Και να σα πω και το εξή ότι σίγουρα ε, ε, είναι σημαντικές αυτές ε, οι συναντήσεις αντιπαράθεσης, διαλόγου. Αν μη τι άλλο, για να γνωρίζουμε όλοι αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη, αυτό το οποίο γίνεται εδώ, αν θέλετε, στις Βρυξέλλες. Γιατί κοιτάξτε, εγώ θα σας το πω χωρί, απερίφραστα. Οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη και τις αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ σαν κάτι το πολύ μακρινό. Αλλά όχι μόνο οι πολίτε. Μερικέ φορέ και τα εθνικά κοινοβούλια και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Θα σα πω το εξή. Άκουσα πριν από λίγο τη Συντόνια, η οποία μιλούσε για ένα εμβληματικό ε, σχέδιο που είχε να κάνει με, τους, ε, με, τις, ε, με τη μετακίνηση των νέων. Εγώ δεν το γνώριζα. Ναι, ενδεχομένως να φταίω εγώ που δεν είχα διαβάσει και δεν είχα ενημερωθεί. Αλλά πόσοι νέοι στην Ευρώπη γνωρίζουν για την ύπαρξη αυτού του προγράμματο που του αφορά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει και το οποίο ε, ε, βρίσκεται ανάμεσα στους πολίτες της Ευρώπης και στην Ευρώπη, δικό μας καθήκον ε, και εδώ πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να καταφέρουν να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο λαό της Ευρώπης και στους ίδιους θεσμούς της Ευρώπης. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου η ευχή και σας, θα ήθελα να σας παροτρύνω να συνεχίσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα λοιπόν ε, Youth in the Move στα αγγλικά, νεολαία σε δράση, ε, είναι πρόσφατο και δεν το γνωρίζουν πολύ ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να σας πω ότι έχετε δίκιο όμως, πέραν τούτου. Ζούμε σε δύο ξεχωριστούς κόσμους και αυτό είναι παράλογο. Τα προβλήματα είναι κοινά. Και οι αρμοδιότητες μας συμπληρώνουν η μία την άλλη. Γύρω στο 2005, ένα μεγάλο υπουργός οικονομικών, μια ημέρα στο Συμβούλιο των Υπουργών, έθεσε το εξή ερώτημα. Ρώτησε ποια, ποια ήταν, πόσοι υπουργοί τη γαλλική κυβέρνηση ήξεραν ε, για τη Λισαβόνα. Που είχε ξεκινήσει το 2000 το πρόγραμμα τη Λισαβόνα. Ε, σα λέω ότι πάνω από το 50% ε, των υπουργών δεν γνώριζε καθόλου το θέμα αυτό. Και κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για του Γάλλου υπουργού. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, τα πράγματα και επειδή δεν ήταν καλύτερε και αλλού. Αν θέλουμε λοιπόν να πετύχει η στρατηγική Ευρώπη 2020, πρέπει να τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, συνδέσουμε και την εθνική κοινή γνώμη. Και αυτό μπορεί να το κάνουν πολύ πιο εύκολα τα εθνικά κοινοβούλια σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε την εξή ιδιαιτερότητα. Κανεί δεν μιλά ποτέ για μα. Αυτή είναι η ιδιομορφία μα. Αυτό είναι και πλεονέκτημα βέβαια. Σε ορισμένες, φορές αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε επίπεδο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής είναι καταστροφή. Γιατί αν δεν μιλάει κανείς για σένα, τότε κανείς δεν σε ξέρει. Ε, αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Ε, όμως ακόμα και ο ειδικό τύπος ε, για τα ευρωπαϊκά θέματα βρίσκεται στο περιθώριο. Θεωρούνται ως εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι και ότι τα θέματα είναι ιδιαίτερα τεχνικά κτλ. Ναι, ε, αυτή είναι η εικόνα και σε, πολλές, ε, και σε πολλά κράτη-μέλη. Μας θεωρούν ειδικού που βρισκόμαστε στο περιθώριο. Κοιτάξτε, στο παρελθόν που οι αρμοδιότητέ μα δεν ήταν μεγάλε, δεν είχε τόση σημασία. Αλλά τώρα με τη Λισαβόνα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ένα λοιπόν από τα ατού που έχουμε είναι να συνδέσουμε ε, τα, τα εθνικά κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Γιατί μέσω των εθνικών κοινοβουλίων έχουμε πρόσβαση στα μέσα μαζική ενημέρωση εθνικό επίπεδο και στου πολίτε σε τελευταία ανάλυση. Γιατί τα εθνικά κοινοβούλια έχουν άμεση σχέση με τους πολίτες σε σχέση με εμάς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκοντμάνης. Ε, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την ε, Λετωνία και έχω πείρα διότι υπήρξα και εγώ υπουργό Οικονομικών. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι η διαφορά είναι τεράστια διότι ε, στο Εθνικό Κοινοβούλιο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όταν δεν υπάρχουν τα αναγκαία έσοδα ενώ εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά έχουμε δεσμεύσεις και πληρωμές ε, που δεν είναι το ίδιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά στο τέλος εάν κοιτάξετε την κατάληξη τον τελικό αριθμό ε, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται έρχεται από τα εθνικά κοινοβούλια. Το, στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι αριθμοί είναι πολύ περιορισμένοι. Αν δείτε λοιπόν το έγγραφο του κυρίου Λαμασούρη η κατάσταση είναι δραματική. Αν ερμηνεύσει κανείς το κείμενο αυτό βλέπουμε ότι αν αναλάβουμε νέες προσκλήσεις, προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την Ευρώπη του 2020 δεν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση γιατί μεγάλη αριθμοί ε, χωρίζονται στα δύο. Αφενός η γεωργία η οποία ε, είναι δεσμευμένη μέχρι το 2013 και δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουμε πολλά και τέλος μέχρι το 2000 μέχρι πρόσφατα τα προγράμματα δεν ήταν έτοιμα οπότε αντί τα χρήματα να, να τεθούν στα αρχικά προγράμματα διετέθησαν στα προγράμματα ανακάμψεως και τώρα λείπουν και το δεύτερο μέρος των δαπανών, τα διαρθρωτικά ταμεία και αυτά ε, είναι δεσμευμένα και λιμένα μέχρι το 2013. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας. Γι' αυτό οι νέες προκλήσεις που αναγράφονται στην ατζέντα του 2020, κλιματολογικές αλλαγές, μετά επανερχόμαστε στις κοινέ εξωτερικές δράσεις κτλ. είναι πολύ προβληματικές διότι τα χρήματα δεν επαρκούν. Και το ερώτημα είναι ή δύο πράγματα. Ή θα πρέπει εσείς να δώσετε περισσότερα χρήματα το οποίο δεν είναι και τόσο δυνατόν διότι οι περισσότεροι από εσά έχετε προβλήματα στον προπολογισμό σας ή θα πρέπει να ανακυκλώσουμε και να διαρθρώσουμε τη χρηματοδότηση εσωτερικά και ορισμένοι θα πρέπει ε, να πάρουν λιγότερο και άλλοι να πληρώσουν περισσότερο. Γι' αυτό και στην αναθεώρηση που θα γίνει στο μέσο της διαδρομής ε, δεν πιστεύω ότι θα έρθουν και θα βρεθούν νέοι πόροι και θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα όπου καταβάλουμε πάρα πολλά. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, αν είστε ικανοποιημένοι τα κοινοβουλιά σας οι εκπρόσωποι του λαού είσαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό και δεν αναφέρομαι μόνο στους, ε, στα μεγάλα κονδύλια αλλά και στις τάσεις Προσπάθησα να κάνω μία ανάλυση από το 2007 ως τον προϋπολογισμό του 2011, δηλαδή μέχρι το σήμερα. Και βλέπω ότι προβλέπουμε το 2011 να πληρώνουμε λιγότερο από το 2007. Και ποια είναι αυτές οι βασικές θέσεις. Είναι επώδυνες ε, στην απασχόληση και κοινωνική ε, ε, ασφάλιση 18% λιγότερο ε, και ο λόγος είναι ότι δεν πληρώσαμε ε, επαρκώς τα, τα κοινωνικά ταμεία στην αρχή μέσω των δεσμεύσεων διότι ναι μεν είχαν ε, προγραμματίσει πολλά τα οποία όμως δεν δώσαμε διότι δεν ήταν έτοιμα τα προγράμματα και τα χρησιμοποίησαμε αλλού και στις παλιές και στις νέες χώρες όταν υπάρχουν τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης ε, ε, δημιουργείται μια φέμαξη των διαρθρωτικών ταμείων και βλέπουμε ότι οι πληρωμές μας είναι τελικά μικρότερες από το 2007 και νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε έλλειψη αποδοτικότητας δηλαδή ε, στην έρευνα οι ε, επιστήμονες δεν μπορούν ε, να μας δώσουν επαρκή ικανοποιητικά προγράμματα για τα ναυτιλιακά πολλοί θα δυσαρεστηθούν 21% λιγότερες πληρωμές από ότι το 2007 γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις διεθνείς συμφωνίες και γι' αυτό το λόγο έχουμε λιγότερες πληρωμές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές θέσεις όπου προσπαθούμε να αυξήσουμε τις καταβολές μας ε, και αυτό δεν αναφέρεται στο έγγραφο του κυρίου Λαμασούρ και είναι ένα θαύμα κατόπιν της κρίσεως το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κατάφεραν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για προγράμματα εθνικής ανακάμψεως. Μπόρεσαν να βρουν πολλά χρήματα και παρόλο που είναι απίστευτο το πρόγραμμα πέτυχε ε, για προγράμματα ε, έρευνας ε, για το Ταμείο Γάλακτος και το καθεξής αλλά αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει μόνο μία φορά όπως σας είπα και από τα διαρθρωτικά ταμεία διότι η εφαρμογή είναι χειρότερη από ό,τι σε προηγούμενες περιόδους Ιδίω ιδίως λόγω της κρίσεως και τώρα προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε και άλλους πόρους. Τελικά υπάρχουν θετικά ε, σημεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε 251% περισσότερα το 2011 από ό,τι πληρώσαμε το 2007. Στις μεταφορές 202% περισσότερα το 2011 σε σχέση με το 2007. Δηλαδή ε, σε αυτές τις ε, ενδιάμεσες περιόδους μπορεί να είχαμε ζημίες αλλά προσπαθούμε ε, να αντιδράσουμε στην κρίση, να αυξήσουμε τις μεταφορές μας και για την έρευνα υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως θα υπάρξουν 59% περισσότερο πληρωμές. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο χρηματοδοτήσαμε στο παρελθόν τον τομέα αυτό ε, τώρα ε, θα προσπαθήσουμε ε, να ισοσκελίσουμε την κατάσταση. Κοιτάξτε λοιπόν τη διαφορά μεταξύ 2011 με 2007 και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουμε διαφορά πληρωμών 67%. Υποθέτω όμως ότι τους λογαριασμούς το κάνει και κάθε κράτος ε, στην αντίστροφη κατά, ε, ε, κατεύθυνση. Προσπαθούμε εμείς να μοιράσουμε κονδύλια ε, ε, μπορεί να είναι 37 εκατομμύρια ε, μόνο περισσότερα αλλά αναλογικά είναι 67% περισσότερα και για την προστασία των καταναλωτών έχουμε διαφορά 107% δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι παραβλέψαμε αυτά τα σημαντικά κοινά θέματα δικαιώματα και ε, έχουμε 655 περισσότερα εκατομμύρια που θα πληρώσουμε για την ασφάλεια το 2011 από το 2007. Δηλαδή έχουμε πάνω από 200% αύξηση. Και όσοι ενδιαφέρονται ε, για την ελευθερία και για αυτά τα θέματα δεν μπορούν να παραπονούνται. Και στο τέλος επανέρχομαι αυτό το οποίο έγραψε ο κύριος Λαμασούρη τουλάχιστον υπονοεί ε, ανάμεσα μέσα στις, ε, στα λόγια του ότι ε, ίσως θα γίνει η αξιολόγηση του, με, ε, στο μέσο της διαδρομής ε, για τον ε, προϋπολογισμό. Δεν έχουμε όμως μέθοδο εδώ. Δεν υπάρχει μία σοβαρή προσέγγιση και δεν νομίζω ότι θα οικονομήσουμε ακόμη πολλά κεφάλαια και θα χρειαστεί να ισοσκελίσουμε. Δηλαδή, αν ανατάξουμε τις πιστώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε διότι το 1% δεν επαρκεί όπως έγραψε ο κύριος Λαμασούρ και αν περιορίσετε λίγο τον προϋπολογισμό της Ευρώπης δεν θα σας συμπαθήσουν ή στα εθνικά σας κοινοβούλια και έχω προσωπική πείρα επ' αυτού. Αλλά με τις συνέργειες μπορούμε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα διότι αν κοιτάξετε τους αριθμούς δεν νομίζω ότι θα επιτύχουμε. Ήταν πολύ βασικό, ε, ε, βασική η συνεδρίαση αυτή. Ε, πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν ήμουν στο Συμβούλιο όταν ξεκίνησε η κρίση και είδα τι γινόταν, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνουν τα κοινοβούλια. Εσείς κρατιάτε τα ενία και άρα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ας παραμείνουμε στη Βαλτική. Ο κύριος Κάρσουλα, εκ μέρους της Κούντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκ μέρους του Φιλανδικού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής των Οικονομικών έχω εγώ προσωπικό τη δυνατότητα να συμμετάσχω στην ε, συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την όλη προσπάθεια της οργάνωσης της συνεδρίασης. Η κρίση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία, υπόθηκε και το πιστεύω και εγώ. Πολλά αντίστοιχα παραδείγματα έχει να επιδείξει η ιστορία. Ο πρόεδρος έδωσε την οικογένεια ως παράδειγμα. Και βλέπουμε, πιστεύω, ότι μερικές φορές οι κρίσεις ενισχύουν και τους δεσμούς και το άτομο μέσα στην οικογένεια. Η ενότητα της Ευρώπης, η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών δεσμών θα κριθεί από τον τρόπο και πάνω απ' όλα από τη διαφάνεια με την οποία θα δράσουμε από εδώ και μπρος. Και έτσι θα ήθελα να πω ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να διατηρήσει ως κύριο χαρακτηριστικό του την διαφάνεια, ως υπόβαθρο της λειτουργίας του την διαφάνεια. Στη Φιλανδία εμείς έχοντας εξετάσει την κατάσταση επιλέξαμε, μάλλον διαπιστώνουμε ότι περάσαμε τα πιο δύσκολα, προχωρούμε προς μια πιο ικανοποιητική ανάπτυξη και βλέπουμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 άρχισε να εισάγεται η έννοια του προϋπολογισμού πλαισίου ή του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, δηλαδή μιας τετραετίας για την οποία προσδιορίζεται ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο σε τελευταία ανάλυση επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία. Και αυτή είναι ακριβώς την σημασία του δημοσιονομικού πλαισίου διαπιστώνουμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό συνεπάγεται και ενισχυμένη συνεργασία. Συνεπάγεται περισσότερη ε, πιο αλληλένδετη δράση και έχει σαν απόρρια περισσότερη εμπιστοσύνη και αποτελεσματικότητα στην χρήση των κεφαλαίων. Ας επανέλθω όμως στην έννοια της εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της ε, εμπιστοσύνης. Να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, ότι εγώ ερχόμενο εδώ σκεφτόμουν ότι θα δω καλούς φίλους, θα συναντήσω γείτονες αγαπητούς και ότι θα έχουμε εδώ στην Ευρώπη μία καλή, αποτελεσματική συνεργασία. Μια συνεργασία η οποία δεν θα διαμορφώνεται μόνο με όρους γραφειοκρατίας αλλά θα αποτελέσει και μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία την οποία θα ενισχύσει και η καινοτομία και ε, θα οδηγήσει σε περισσότερη ευημερία. Και γι' αυτό θα μπορέσει η Ευρώπη να καταστεί πρωτοπόρος. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σχέση μεταξύ του Εθνικού, των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο, ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουμε και για την περαιτέρω συνεργασία μα. γιατί πρέπει πάντα να κοιτάμε προς τα μπρο και γι' αυτό, Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα του πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τις περαιτέρω σχέσεις, τις εξελίξεις Πρόκειται για ένα ερώτημα κλειδί πιστεύω. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις εξελίξεις, πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μία αηφόρο οικονομία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη επιμέρους και εδώ θα ήθελα να πω εγώ ότι η συνθήκη της Λισαβόνας και η στράτευση την οποία ε, αναλαμβάνουμε ίσως απαιτεί περισσότερη αποφασιστικότητα από τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι πρέπει περισσότερο να ασχοληθούμε, να επικεντρωθούμε στο ερώτημα του πώς η Ευρώπη του 2020, η στρατηγική αυτή ενισχύεται, θα ενισχυθεί και στο εθνικό επίπεδο και μέσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, πώς θα τις προσδώσουμε ουσία. Πώς τα κράτη-μέλη θα επιτελέσουν το καθήκον που έχουν, έχουν με την διαδικασία της Λισαβόνας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, μια διάσταση μάλλον πιο επίσης σημαντική, είναι το δημοκρατικό έλλειμμα. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων, δημοκρατικός τρόπος λήψης αποφάσεων και η αναφορά στο διεθνές πλαίσιο ή στην παγκοσμιοποίηση. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ασφαλώς κοινός διάλογος θα είναι χρήσιμη η συζήτηση του πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατική διάσταση, πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα. Το Youth on the Move, νεολαία εν κινήσει, είναι μια πολύ καλή προοπτική για το 2020, ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ένα σημείο στο οποίο έχουμε, πιστεύω, ουσιαστική απεικόνηση της προσφοράς που μπορεί να σημάνει η Ευρώπη. Όταν δηλαδή οι νέοι μας μπορούν να ε, επισκέπτονται ο ένας τον άλλον, να έχουν ελεύθερη διακίνηση, να γνωρίζουν ε, τον ένα και τον άλλο τόπο, κερδίζουμε όλοι, κερδίζει όλη η Ευρώπη. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας, ετέρα τη Φινλανδία, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε δει σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας ότι οι νέοι όπου ταξίδεψαν, όπου επισκέφτηκαν, όπου αποκόμισαν νέες παραστάσεις και ιδέες, μπόρεσαν να προσφέρουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να το δούμε πιστεύω και με την ε, και υπό τη σκιά ίσως της ε, ανεργίας των νέων, μιας μεγάλης πρόκλησης την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, την οποία θα πρέπει πιστεύω να λύσουμε ενισχύοντας το επιχειρηματικό πνεύμα. Και Πρόεδρε πιστεύω ότι ακόμη και αυτές οι συζητήσεις, οι δικές μας οι συναντήσεις, οι διασκέψεις μπορούν να ε, οργανωθούν στο μέλλον σε πιο συγκεκριμένα θέματα, να επικεντρωνόμαστε δηλαδή σε μια συγκεκριμένη θεματολογία και να ε, προσδορίσουμε έτσι και τους εθνικούς προπολογισμού με περισσότερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και πολλά διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε από την εμπειρία της Φιλανδίας. Είχα την τιμή να συμμετάσχω στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην ένταξη της Φιλανδίας μαζί με τη Σουηδία και την Αυστρία πριν από 15 χρόνια και τότε η οικονομική κατάσταση στη χώρα σας ήταν καταστροφική γιατί έπρεπε να αλλάξετε τελείως τον προσανατολισμό της οικονομίας σας που μέχρι τότε ήταν στραμμένη προς τη Σοβιετική Ένωση και έπρεπε να την στρέψετε προς την Ευρωπαϊκή ε, ήταν στραμμένη προ τη Σοβιετική Ένωση και έπρεπε τώρα στην προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απέτυσε πολλέ θυσίε και αποτελέσματα μέσα σε λίγα χρόνια. Μα αυτά όμω είναι και καλά νέα, γιατί σημαίνει ότι όλοι, αν δείξουμε το ίδιο θάρρο και ασκήσουμε τι ίδιε προσπάθειε, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Ε, ε όσον αφορά τι επιδόσει σα στην εκπαίδευση, και έχουμε αποτύχει σε πολλέ χώρε εμεί στον τομέα τη παιδεία, δυστυχώ και στη χώρα μου. Και όμω εσεί είσαστε παράδειγμα ε, σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα τη παιδεία. Και επίση. Ε, ε, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προβλήματα και την ε, οργάνωσή σας ε, σε επίπεδο κοινοβουλίου της χώρας σας που έχετε φτιάξει αυτή την επιτροπή και ε, μπορούν με αυτόν τον τρόπο όλοι οι πρωτοβουλίε του Φινλανδικού Κοινοβουλίου να συνδέονται με τον έλεγχο της ευρωπαϊκής πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνησή σας. Πραγματικά έχετε να μας προσφέρετε πολλά παραδείγματα. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στα τρομερά προβλήματα που δημιουργούνται και σε δημοσιονομικό επίπεδο λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Ε, πρόβλημα χρηματοδότησης των συντάξεων, πρόβλημα περίθαλψης, χρηματοδότησης της ε, περίθαλψης του γυράσκοντος πληθυσμού. Και θα έλεγα ότι υπάρχουν προβλήματα που είναι λιγότερο ορατά και που αφήν, αφορούν την έλλειψη, την απώλεια δυναμισμού το τόνισαν ιδιαίτερα ορισμένες, ευρωπαϊκέ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που μίλησαν ε, για χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στο ότι η φυσική δυναμική ε, που προσδίδουν ε, οι πολλοί νέοι σε μια χώρα εδώ έχουμε αυτά τα προβλήματα. Και σας παραθέτω το παράδειγμα της Ιαπωνίας. Εδώ και 15 χρόνια η Ιαπωνία αντιμετωπίζει μια κρίση και δεν μπορεί να φύγει από αυτή την κρίση. Μα είναι μια χώρα με πληθυσμό που γερνάει. Απ' την άλλη έχουμε παραδείγματα χωρών που επιτυγχάνουν όπως ε, η Φινλανδία. Έχουμε λοιπόν πολλά πρότυπα. Ε, τώρα, να δώσουμε το λόγο στους τελευταίους ομιλητές, τον κύριο Φερνάντ ε, που εκπροσωπεί το ΕΛΚ σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εξαιρετική ποιότητα των, της σημερινής μας συζήτησης. Επίση, ε, θα ήθελα να πω ότι το έγγραφο εργασία είναι ιδιαίτερα καλό και εκφράζουμε την ικανοποίησή μα ε, για την ικανοποίηση αυτή. Επί τη ουσία, μιλάμε για την ενίσχυση τη δημοκρατική νομιμότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα Ε, φροντίζει έτσι ώστε ε, προσπαθεί να ακουστεί η φωνή του. Και δεν το πετύχαμε πάντα. Ε, θέλουμε τώρα λίγο περισσότερο. Και αυτό πιστεύω ότι ε, θα επιτευχθεί και με την περισσότερη ολοκλήρωση. Γιατί αυτό, ε, θα, αυτό θέλουν οι πολίτε οι οποίοι αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται καλύτερα από τα κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ολοκλήρωση. Και αυτή η περισσότερη ολοκλήρωση και η περισσότερη Ευρώπη θα, συνε... θα προσδώσει ε, και περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία. Άκουσα ε, διάφορα ζητήματα να αναφέρονται και άκουσα επίσης ε, ε, την καταπολέμηση ε, των απατών και, την, και τον, τον έλεγχο. Ναι, ναι, βεβαίως, έλεγχος και επαγρύπνηση. Που, και, και θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και σαφήνεια σε αυτό το μηχανισμό εποπτείας και πρόληψης. Μιλώ για τα ελλείμματα. Αυτό Κοιτάξτε, ε, και ε, πιστεύω ότι εδώ, σε αυτή τη δικασία θα πρέπει να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις κυρώσεις, εδώ πρέπει να δούμε τους πολίτες. Επιβολή διπλής τιμωρίας, αν θέλετε. Ε, οι εθνικέ κυβερνήσει τιμωρούν τους πολίτες και τους ζητούν να σφίξουν το ζωνάρι μέσα από προγράμματα λιτότητα. Θα του επιβάλλουμε λοιπόν διπλή ποινή. οι πολίτες φταίνε μόνο γιατί επέλεξαν αυτές τις ανίκανε κυβερνήσεις. Επίση, αναφέρθηκε η ανάγκη να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Όσον αφορά τα προγράμματά μας, ε, ε, τον προπολογισμό μας. Ναι, να σας πω το εξή. Όσον αφορά τα, τα χρήματα τα οποία δεν δαπανώνται σε αιτήσιο επίπεδο, νομίζω ότι θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο ή, και γιατί όχι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του προπολογισμού του επόμενου έτους. Το 2001 είχαμε ένα πλεόνασμα ε, σημαντικό και δεν αξιοποιήσαμε τα χρήματα αυτά για την ενίσχυση του επόμενου προπολογισμού ή για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής για παράδειγμα, την καταπολέμηση φτώχειας κτλ. Δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να ε, προωθήσουμε περισσότερο τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ταυτόχρονα πιστεύω θα ήταν σωστό και το λέω τώρα που έχουμε και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να σκεφτούμε και την δυνατότητα και την πιθανότητα να έχουμε επενδυτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόθεση της κινητικότητας αν θέλετε. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε του εθνικού προπολογισμού με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να, να πω ότι ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία αυτή, για το έγγραφο εργασία και για αυτή την ε, ανάγκη ενίσχυση τη νομιμότητα για να μπορέσουμε να δράσουμε με πολύ πιο σωστό τρόπο. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την διοργάνωση αυτή. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Τελευταίο ομιλητή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο οποίο και θα λάβει τελευταίο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα πολλά να πω, αλλά απογοητεύτηκα διότι δεν υπάρχει εδώ κανείς εκπρόσωπος του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω εάν αυτό οφείλεται ή στο νέο Κοινοβούλιο ή στη νέα κυβέρνηση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ε, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την Ουαλία ή μια άλλη περιοχή όπου θα είχαμε πιο θετική ε, απάντηση από από το ε, Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, ε, ε, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δημοφιλές στην Αγγλία το θέμα του συντονισμού του Ευρωπαϊκού ε, Προϋπολογισμού με ε, τον Βρετανικό. Υπάρχουν διάφοροι σκεπτικιστές οι οποίοι απαιτούν λιγότερο συντονισμό και λιγότερη χρηματοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι ήδη στόχοι με αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει αυτό να το αναφέρουμε. Ε, δηλαδή υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία είναι πολύ βασικό θέμα για να υπάρχει καλή, καλό συντονισμός μεταξύ Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων και θα πρέπει τα διαρθρωτικά ταμεία να έχουν επαρκή χρηματοδότηση ε, ε, αλλά πρέπει να πούμε ότι πέραν αυτού του θέματος το οποίο ίσως είναι της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν την ε, κατάσταση ε, για να φροντίζουν για την ευημερία και τα ωφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι πολίτες της Ευρώπης όπως άλλωστε και από το θέμα της ε, ε, ε, γεωργικής πολιτικής. Σήμερα μιλήσαμε για τους πόρους, αλλά νομίζω ότι οι ευκαιρίες σαν τη σημερινή πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον για συζήτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, για χρηματοδότηση των μικρών ε, επιχειρήσεων οι οποίες ε, θέλουν να διευρυθούν και χρειάζονται ένα ταμείο αναζωογονήσεως κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές ευκαιρίες να εμπλακούν τα εθνικά κοινοβούλια για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά τρόπον ώστε η τράπεζα αυτή να έχει τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσει να λειτουργήσει ορθά και ε, είναι θέματα τα οποία ούτως ή άλλως μετακυλούν. Δηλαδή αν υπάρχει στενότητα σε εθνικό επίπεδο μεταφέρεται και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν νομίζω ότι είναι προς όφελος κανενός. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε εδώ και μπορώ να διατυπώσω τα συμπεράσματα των εργασιών. Συντόνια, θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα σας κρατήσω. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα 15 λεπτά που ορίζει η σε διάταξη. Μπορώ πολύ σύντομα, νομίζω, να συνοψίσω αυτή την ανταλλαγή απόψεων ως εξής. ή μάλλον να πω ότι δεν είμαι σε θέση να συνοψίσω, αλλά καθίσταται πιστεύω σαφές από τα όσα ακούστηκαν, ότι όλοι θέλουν να συνεχιστεί ο διάλογος. Όπως αυτός κρίνεται σημαντικός, πρόκειται το διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο ο ευρωπαϊκός και οι εθνικοί προϋπολογισμοί μπορούν να έχουν συμπληρωματική δράση ε, διάλογος για τη σύμπραξη, στην οποία αναφερθήκαμε, και διάλογος ο οποίος είναι χρήσιμος, διότι το να εργαζόμαστε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, εμείς οι Ευρωβουλευτές, φέρνει την πρόσθετη διάσταση, διότι ναι μεν υπάρχουν οι βουλευτές οι οποίοι είναι στις ε, ε, επιτροπέ ευρωπαϊκών θεμάτων των Εθνικών Κοινοβουλίων συνήθω σε επαφή μαζί μα, αλλά δεν βλέπουμε πολύ συχνά συναδέλφου από τι αντίστοιχε επιτροπέ προπολογισμών ή οικονομία κτλ. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο, μια παράμετρο η οποία πιστεύω ανοίγει του οριζοντέ μα, μα επιτρέπει να έχουμε επικοινωνία σε θέματα ε, προπολογισμών, γιατί μέχρι τώρα είμαστε μόνο περιορισμένοι εμεί από την Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου σε επικοινωνία με του υπουργού του αρμόδιου. Ε, και επίσης δεν ήθελα να πω, ε, υπενθυμίζοντας τα όσα στο ψηφισμά του του Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, ότι την πορεία για το 2020 θα πρέπει να τη με γνώμονα την νεολαία. Με σοβαρότητα και με ευθύνη πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για την νεολαία, για τη μόρφωσή της, για την επιμόρφωσή της, για την κινητικότητα. Γιατί οι νέοι είναι, θα έλεγα, φυσικός σπόρος για την Ευρώπη και μάλιστα φυσικός σπόρος που θέλει να εκλείψει. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε πιστεύω όλοι, αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη όλοι. Και μάλιστα ε, θα επισημάνω ότι πρόκειται για την ε, ίσως λιγότερο δαπανηρή, την πιο φθηνή και ίσως και την πιο αποδοτική επένδυση για το μέλλον. Η επένδυση που θα κάνουμε στους νέους μας, στην νεολαία μας. Επίσης, σημειώνω ότι δεν ε, μπορεί να αποφευθεί συζήτηση σχετική με την ευρύτερη μακροοικονομική κατάσταση, το υπόβαθρο δηλαδή της κρίσης που έχει ανασκέψει στην Ευρώπη και συμφωνώ με την ιδέα που ακούστηκε νωρίτερα ότι κατά παράδοξο τρόπο η όλο και πιο αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, η αποταμίευση προς η, οικονομία στους πόρους καλύτερα, ενισχύει την κοινοτική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν την κρίση αυτή θα πρέπει να τη δούμε ως μια ευκαιρία και πολλοί ε, συνάδελφοι ε, διατύπωσαν ενδιαφέροντα παραδείγματα, ένα από αυτά ήταν της Φιλανδίας, που πιστεύω μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να διδαχθούμε από αυτά και χάρη σε αυτά να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά προς το μέλλον. Επισημένω δε ότι έχουμε τρεις νέες υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών στο μέλλον και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο επίλυσης των προβλημάτων και κριτικής εξέτασης των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε. Ακούστηκαν διάφορες ιδέες για το πρόγραμμα για το 2020 και τις βασικές ιδέες ε, που διατυπώνουμε. Ιδέες που μερικές φορές υπάρχουν ήδη αλλά προσλαμβάνουν νέα, νέους τίτλους. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας, θα μας υποστηρίξει στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε προγράμματα που υπάρχουν ήδη και που έχουν φέρει καρπούς όπως το Youth in Action, η, η διαβίου, μάθηση, ε, με το ονομαζόμενα ίσως διατηρούν τους πόρους τους και από την άλλη πλευρά να ε, προχωρήσουμε στην ανάπτυξη νέων σχεδίων, νέων προγραμμάτων με την προοπτική του 2020. Στόχος μας νομίζω θα πρέπει να είναι και να διαφυλάξουμε τους δικαιούχους που ήδη έχουν ε, αποδείξει ικανότητες και αποτελεσματικότητα και να προχωρήσουμε προς νέες λύσεις χωρίς να ανατρέπουμε τίποτα. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι βλέπω αυτή μας τη συνάντηση ως μια απαρχή διαλόγου και ελπίζω οι νέες εξουσίες που απορρέουν από το πρωτόκολλο της συνθήκης, προσάρτημα της συνθήκης Λισαβόνας να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε με έγκαιρη επικοινωνία διάλογο και ταυτόχρονα διάκριση της ευρωπαϊκής από την εθνική διάσταση, διαφυλάσσοντας τις εθνικές εξουσίες και προνομίες, αλλά ταυτόχρονα και συντονίζοντας τις δραστηριότητες μας από το ευρωπαϊκό και το εθνικό ε, επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Συντόνια. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στις ε, συζητήσεις μας σήμερα. Πιστεύω ότι όλοι ιδιαίτερως ε, εκτιμούν τις προσπάθειες και το έργο της Συντόνια, τα όσα μας είπε. Ευχαριστούμε όλους που ήταν παρόντας εδώ και έλαβαν μέρος στις συζητήσεις. Εγώ καταγράφω και σημειώνω την ίσως κάπως προκλητική διατύπωση του Γκόραν Φέρμ νωρίτερα ότι είναι, ε, έχουμε περιέλθει σε κρίση, ας μην χάσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο μήνυμα που πρέπει να αποκομίσουμε από αυτήν την κατάσταση. Και θα υπενθυμίσω και μια παρατήρηση του Τσέρτσιλ, μια κουβέντα που είχε πει για του Αμερικανού. Είχε πει λοιπόν ο Τσέρτσιλ ότι οι Αμερικανοί, έχοντα ε, ε, δοκιμάσει κάθε πιθανή λύση, καταλήγουν πάντα στην καλύτερη. Εν τέλει, περί πρόκειται βέβαια. Για εμά, δεν του Γάλλου, που τουλάχιστον στα δημοσιονομικά εδώ και 20 χρόνια να ζητούμε την καλή λύση και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει. Ε, θα σημειώσω ότι μάλλον δεν θα τη βρούμε την καλή λύση. Γιατί, Γιατί ψάχνουμε μόνο χαλική λύση και δεν κοιτάμε πώ έχει κανεί άλλο πριν από εμά εφεύρει τον τροχό. Εμεί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα τροχό που θα είναι τετράγωνο. Ε, ίσως λοιπόν να δούμε, να δούμε όλοι, όχι μόνο εμείς οι Γάλλοι, ότι κάπου σε έναν άλλο τομέα ένας εταίρος έχει πριν από μας εφεύρει τον τροχό του 21ου αιώνα. Και προσωπικώς από τη συζήτηση κρατώ το εξής, ότι η ιδιαίτερη συνένεση διατυπώνεται από όλους τους ομιλητές ως προς την ιδέα να γίνεται κάθε χρόνο μια κοινή συνάντηση, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αυτή να είναι η αρχή, μια συνάντηση για τον προϋπολογισμό. Επαναλαμβάνω, Βέβαια, ο κάθε ένας από τους εδώ ε, παρόντες μίλησε μόνο προσωπικά, δεν δεσμεύει και δεν εκπροσωπεί με τις δηλώσεις του κανένα ε, κράτος μέλος. Ε, μάλιστα, από τους Γάλλους συναδέλφους θα πρέπει να πω ότι ανήκουν στην αντιπολίτευση, Επομένω, δεν εκφράζουν τις θέσεις της κυβέρνησης. Αλλά τουλάχιστον ξεκινούμε με αυτές τις θέσεις και τις προβάλλουμε. Και επίσης σημειώνω ότι εκφράστηκε ευρύτερη υποστήριξη στην ιδέα να συνεχίσουμε τη συνεργασία για να επιβάλλουμε τις προνομίες των κοινοβουλίων και να ασκήσουμε το λειτουργήμα του κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων μέσα στην ε, δημοκρατική λειτουργία και την εφαρμογή βέβαια των δραστηριοτήτων, ε, των οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάπτυξη δηλαδή που χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερος δε ε, σημειώνω ότι εάν να εξασφαλίσουμε αυτή την ετήσια ε, διάσκεψη για τα δημοσιονομικά με συμμετοχή και των κρατών μαλλών, τουλάχιστον τριών ειδών θέματα θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστούν. Συντονισμός δημοσιονομικός, αυτός καθεαυτός που υπόθηκε νωρίτερα, που αναφέρθηκε πολλές φορές μάλιστα. Ε, εξέταση και αντιμετώπιση των λεγόμενων κρίζων, γκρίζων ζωνών ή των παραθυρακίων, όπως υπόθηκε νωρίτερα από τον συνάδελφο το Γάρλο, ε, δηλαδή τις αποφάσεις που λαμβάνουν μένει οι θύνοντες, οι οποίες όμως ε, διαφεύγουν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αλλά και του Εθνικού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου γιατί όταν ξεκίνησε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, η μεγάλη τραπεζική κρίση καλύτερα ε, διατυπώθηκε η κατηγορία ότι δεν υπήρχε εξέταση του μεγάλου περιθωρίου κέρδους των τραπεζών, των δεσμεύσεων έξω από τον ισολογισμό και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα κράτη-μέλη, δηλαδή για τις δεσμεύσεις που λαμβάνουν έξω από τον προϋπολογισμό. Και έτσι θα πρέπει με αυτό τον τρόπο παρεμβάσεως ελέγχου, κοινοβουλευτικού ελέγχου, να θέσουμε τέρμα σε αυτές τις γκρίζες ζώνες. πολλοί μάλιστα από τους συναδέλφους, αναφέρθηκαν στο ζήτημα των κυρώσεων. Ένα ακαθόδε ζήτημα, ένα ζήτημα για το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί ικανοποιητική λύση. Γιατί βέβαια ο αντιλαμβάνεται ότι αν δεν υπάρχει η έννοια της αποτροπής, ο κίνδυνος, ο οποίος, η απειλή μάλλον η οποία θα αποτρέψει μια χώρα από την κακό διαχείριση, έχουμε πάλι φαινόμενο σε αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Άρα χρειάζεται κάποια αποτροπή. Από την άλλη, η κύρωση που προβλέπεται σήμερα από τις συνθήκες, δηλαδή το να υποβληθεί η χώρα που δεν τηρεί τα όρους του Μαστρίχτ του Συμφωνού Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε δημοσιονομική εποπτεία, επιτήρηση, είναι μάλλον παράλογη κύρωσε, Όπως πόθηκε και νωρίτερα, γιατί απλώς ε, καταστρέφει ένα κράτο ήδη χρεοκοπημένο. Άρα χρειάζεται άλλο μηχανισμό Και πάντως χρειάζεται το θέμα να μην το κοιτάμε μόνο με γνώμονα τις κυρώσει. Όπως λέμε καρότο και, ε, και μπαστούνι, ε, όπως λέμε δούνε και λαβίν, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, και τιμώρησης αλλά και ανταμοιβή ή κινήτρων στις δημοσιονομικές μας μεταρρυθμίσεις και μάλιστα θα θέλω να επενθυμίσω τους ταλού ε, συναδέλφους οι οποίοι όπως και άλλοι μίλησαν και είπαν ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν θα είναι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά αλλά και πρακτικά Σήμερα είδαμε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να έρθουν διότι τα κοινοβούλια δουλεύουν ανά τον κόσμο συνήθω τρίτε τετάρτε, πέμπτες. Και το Σαββατοκύριακο επιστρέφει κανεί στην εκλογική του περιφέρεια για να συναντήσει του ψηφοφόρου του. Άρα η Τρίτη δεν είναι πάντοτε η καλύτερη μέρα για να εξασφαλιστεί η αθρώα προσέλευση των εκπροσώπων των Επιτροπών Προπολογισμών των Κρατών Μελών, των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Θα πρέπει να βρούμε ίσω κάποια άλλη πρακτική λύση. Εγώ θα πρότεινα, σε συνεργασία με τι αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βέβαια με την ε, μελλοντική Βελγική Προεδρία, να δούμε εάν μπορούμε να ε, στήσουμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα μπορούσε να εξετάσει ακριβώς το θέμα της ε, πρακτικής οργάνωσης και της επιλογής συγκεκριμένη μορφής και ημέρας διεξαγωγής μιας πρώτης δημοσιονομικής διάσκεψης, εάν τα καταφέρουμε τελικά. Και προσθέτω, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φαν Ρόμποϊ έχει επιφορτιστεί με την ε, μελέτη της ε, θέσπισης μιας νέας διαδικασίας και νέου μηχανισμού συντονισμού των πολιτικών, οικονομικών πολιτικών και έχει συστήσει ομάδα εργασίας η οποία θα καταθέσει πόρισμα και προτάσει στα τέλη τον ε, του καλοκαιριού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε αυτές τις εργασίες. Η ακριβής μορφή συμμετοχής, διατυπώσεις δηλαδή συμμετοχή ακόμη δεν έχουν προσδοριστεί. Δεν ξέρω εάν τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ζητήσει να παρέμβουν σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, εγώ προσωπικώς, εάν ε, πράγματι ευοδοθεί αυτή η προοπτική, είμαι ε, διατεθειμένος να μεταφέρω τα όσα συζητήθηκαν σήμερα προσωπώντας τους εδώ παρισταμένους αφού ο κύριος Φανρόμποϊ έχει εκδηλώσει βούληση για ε, να ανοίξει τις θύρες πλήρου συμμετοχή στο κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ όλους. Θα κηρύξω το πέρας της σας και σας καλώ, εάν δεν έχετε άλλη δέσμευση, αν δεν είστε υποχρεωμένοι να προλάβετε κάποιο τρένο ή αεροπλάνο, να έρθετε να πιούμε ένα ποτηράκι στο όνομα της φιλίας, στην αίθουσα, εδώ απέναντι, στα αριστερά μας συγκεκριμένα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε πιο οικείο πνεύμα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ.